Bene. Eh. Καλώς. Σας καλωσορίζω όλους αγαπητοί συνάδελφοι. Καλωσορίζουμε και την κυρία Ροκπίλερ η οποία μαζί με την κυρία Κρέτσου θα συμπροεδρεύσει στην ε, σημερινή συνεδρίαση. Ε, έχουμε λοιπόν τον πρόεδρο της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ανάπτυξης που μαζί με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων βρίσκονται εδώ σήμερα για αυτή τη σημαντική ετήσια συνάντησή μας, την παρουσίαση των υποψηφιωτήτων του βραβείου Ζαχάροφ. Από το 1988, πάνω από 20 χρόνια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει αυτή τη σημαντική αναγνώριση σε ανθρώπους και οργανώσεις που απέδειξαν μέσω της δέσμευσή τους, ε, των σκέψεών τους, των δράσεών τους, την ανάγκη ε, η οποία είναι κοινό στόχος της προστασίας των ανθρωπίνων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και ίσως αυτή είναι η πιο συμβολική και πιο αντιπροσωπευτική ένδειξη του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει το Κοινοβούλιο και οι αρχές της ελευθερίας μας. Εμείς ως εκπρόσωποι των πολιτών της Ευρώπης πιστεύουμε στις αξίες που αντιπροσωπεύονται στο βραβείο αυτό. Υποστηρίζουμε την ελευθερία της σκέψης και του λόγου, την καταπολέμηση όλων των ε, παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ελευθερία του τύπου, τη μυσαλλοδοξία, το μίσος, που πολλές φορές συχνά μένουν ατιμέωρητα ε, σε πάρα πολλές περιοχές του κόσμου. Καθήκον μας λοιπόν τις επόμενες ημέρες είναι να βρούμε ποιοι είναι οι άξιοι υποψήφοι για να ξεκινήσει η διαδικασία της λήψης απόφασης η οποία θα επιβεβαιωθεί με την τελική απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων ε, των πολιτικών ομάδων ε, η οποία θα ληφθεί στις 27 Οκτωβρίου όπως γνωρίζετε. Εδώ λοιπόν τελείωσε το δικό μου καλωσόρισμα να δώσουμε λοιπόν το λόγο στην κυρία Λοκμπίλερ, πρόεδρο της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που είναι μια επιτροπή που διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο για την απονομή του βραβείου. Και στη συνέχεια, ε, αφού προεδρεύσει η κυρία Ροκμπίλεν, θα κάνει τις τελικές ε, παρατηρήσεις της η κυρία Κρέτσου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε τώρα παρουσίαση των υποψηφιωτήτων για το βραβείο Ζαχάρο. Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιωτήτων ήταν 14 Σεπτεμβρίου. Έλαβε η Γραμματεία 5 υποψηφιότητες. Η Γραμματεία θεωρεί όλες τις υποψηφιότητες δεκτές στο πλαίσιο του καταστατικού του βραβείου και θα βρείτε στο φάκελό σας ε, σύντομα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων. Έχουμε λοιπόν τον Ισέλτιν Αμπουέλιας, έναν Παλαιστίνιο γιατρό και ιδρυτή του Ιδρύματος ε, Κόρες της Ζωής, ε, τον Ahmed Al Sanusi from Libya, Rasan Saitouni and Ali both from Syria, on behalf of the Arabs. Από την Αραβική Άνοιξη θα λέγαμε κατόπιν Έχουμε τον Δημήτρη Μπανταρέγκα, έναν ακτιβιστή και δημοσιογράφο Λεύκο Ρώσο, Μπόρις Παχόρ, έναν Σλοβένο συγγραφέα πρευστή των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, την ε, κοινότητα του Σαν Χωσέδε Απαρτάδο, μια ειρηνική κοινότητα στην Κολομβία που είναι γνωστή για το ότι υπερασπίζεται τις αξίες της ειρήνης ε, και της δικαιοσύνης. Θα ακούσουμε τώρα τις ε, παρουσιάσεις των υποψηφίων από αυτούς που τους πρότειναν, που θα τονίσουν τα επιτεύγματά τους στους διάφορους τομείς ε, δραστηριοτήτων και στο πολιτικό πλαίσιο. Θα γίνουν λοιπόν ε, οι παρατηρήσεις με αλφαβητική σειρά. Καμιά φορά υπάρχει ένας ομιλητής, άλλες φορές ε, θα μοιράσετε τον χρόνο μιλίας, αλλά δεν θα πρέπει να μιλήσετε για πάνω από 5 λεπτά. Επίσης, η κοινή υποψηφιότητα για την Αραβική Άνοιξη θα έχει 5 λεπτά για κάθε μία από την πολιτική ομάδα που το υποβάλλει και σας παρακαλώ να τηρήσετε το χρόνο. Αν μιλήσετε περισσότερο δεν είναι καλύτερη η παρουσίαση. Στο ζουμί, παρακαλώ. Κάποιες παρουσιάσεις επίσης θα δείξουν βίντεο το πλαίσιο αυτού του πενταλέπτου. Λάβαμε αιτήματα να δείξει βίντεο η ομάδα των ε, Ευρωπαίων Συντητικών και Μεταρρυθμιστών και η ΓΚΟΕ. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τις παρουσιάσεις. Πρώτα απ' όλα θα δώσω τον λόγο στον κύριο Σιέντ Καμάλ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε χρόνο να παρουσιάσουμε τον υποψηφιό μας, τον ε, δόκτωρα Ιζελντίν Αμπουελέης. Γιατί προτείνουμε τον ε, κύριο Αμπολαής είναι λόγω της ε, κατάστασης που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών και βεβαίως αντιλαμβάνομαι και τις υπόλοιπες υποψηφιότητες και εγώ είχα πάει στην Αίγυπτο τον Ιούλιο και δίδασκα τους νέους ακτιβιστές για την ελευθερία, τη δημοκρατία και την ανοχή, είναι σημαντικό να στείλουμε ένα μήνυμα στις δύσκολες αυτές διαπραγματεύσεις πως αντί για πόλωση, αντί να βλέπουμε τη συζήτηση αυτή ότι κάποιος είναι είτε με τους Ισραηλινούς είτε με τους ε, Παλαιστίνιους και εναντίον του άλλου, χρειαζόμαστε ανθρώπους οι οποίοι γεφυρώνουν ε, αυτό το κενό. Εξάλλου, όπως είχε πει και ο Μωσέντα Γιάν, Εάν ε, θέλουμε ειρήνη, δεν μιλάμε στους φίλους μας, μιλάμε στους εχθρούς μας. Και νομίζω πως κανένας άλλος δεν το συμβολίζει αυτό περισσότερο από τον ε, υποψήφιο μας σήμερα. Είναι Παλαιστίνιος γιατρός και ίδρυσε το Ίδρυμα Κόρες για την Ζωή. Σε ολόκληρη την ε, ιατρική του σταδιοδρομία εργάστηκε και σε Παλαιστινιακά νοσοκομεία και με Ισραηλινού ασθενεί. Μεγάλωσε σε στρατόπεδο προσφύγων στη Λωρίδα τη Γάζα. ξεπέρασε πάρα πολλέ δυσκολίε για να γίνει ένα πάρα πολύ αγαπητό ερευνητή και ομιλητή για την ανάπτυξη και την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Αυτό το οποίο ιδιαίτερα μας εμπνέει στον υποψήφιο αυτόν είναι πως ο Δ. Αμπολαής έχασε τρεις κόρες από μια Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση. Σκεφτείτε το, αν έχανε κανείς τα παιδιά μας ή οποιοδήποτε μέλο τη οικογένεια μας πώ αντιδρούσαμε. Νομίζω το ένστικτό μας θα ήταν να μισούμε αυτούς που θα είχαν κάνει αυτό το πράγμα. Και βεβαίως ε, δεν μας αρέσει η λέξη μίσος, αλλά το αντιλαμβάνεται κανείς ε, ε, σε αυτή την περίπτωση ένα τέτοιο συνέστημα. Ανταυτού, σε αυτή την περίπτωση, έχοντα χάσει τι τρει κόρε του, ανταυτού φρόντισε να προωθήσει την ειρήνη, ίδρυσε το Ίδρυμα κόρες για την ειρήνη που σκοπεύει να εκπαιδεύσει του ανθρώπου σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και να ενθαρρύνει ιδιαίτερα την εκπαίδευση των γυναικών. Όχι μόνο των Παλαιστινίων γυναικών και των Ισραηλινών από οπουδήποτε και αν προέρχονται. Αυτά... Αυτό έγινε τον Ιανουάριο του 2009 και έχει συνεχίσει να εμπνέει. Έγραψε ένα βιβλίο που λέγεται «Δεν θα μισήσω» και αναφέρει την ιστορία της ε, ζωής του. Γιατί τον πρότεινα, γιατί θεωρώ πως αυτή τη στιγμή που βλέπουμε πως ε, υπάρχει συζήτηση στον ΟΗΕ για την ανεξαρτησία της Παλαιστίνης, όταν μιλάμε με τους διαπραγματευτές των δύο πλευρών και λένε πως δεν έχουμε συνομιλητή ή δεν μπορούμε να έχουμε λογική συζήτηση με τους διαπραγματευτές της άλλης πλευράς, είναι σημαντικό να κλείσει αυτό το κενό. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στο μίσος να επεκτείνει αυτό το κενό μεταξύ των δύο πλευρών. Ελπίζω με την υποψηφιότητα του Δ. Ιζελντή να μπορέσει να στείλουμε ένα μήνυμα ενθάρρυνση σε Παλαιστινίους και Ισραηλινούς να ξεπεράσουν την εχθρότητα και να συνεργαστούν για την ειρήνη. Ευχαριστώ. Very Σας ευχαριστούμε κυρία Καμάλα. Τώρα για την κοινή υποψηφιότητα της Αραβικής Άνοιξης, εδώ έχουμε διαφόρους συναδέλφους που θέλουν να μιλήσουν. Η κυρία Σαΐφη θα αρχίσει. Merci, Madame la Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι για να χαιρετήσουμε το κουράγιο, την αξιοπρέπεια και την ε, προσήλωση και αποφασιστικότητα των αραβικών λαών που αγωνίστηκαν επί σειρά ετών. Θέλουμε να τιμήσουμε κάποιου από του πρωταγωνιστέ τη Αραβική Άνοιξη. Η απονομή του βραβείου Ζαχάρου φέτο θα λάβει χώρα στι 14 Δεκεμβρίου, το Δεκέμβριο. là, Με ακούτε? Ωραία στις 14 Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο, δηλαδή ένα χρόνο ακριβώς μετά την έναρξη των λαϊκών εξεγέσεων της Αραβικής Άνοιξης. Και πόσο δρόμο κάναμε τον τελευταίο χρόνο. Η δύναμη και η ε, προσήλωσή τους μας ξάφνιασαν και πρέπει να το αναγνωρίσουμε ότι δεν είχαμε αντιληφθεί σε ποιο βαθμό αυτή η δίψα για τη δημοκρατία και την ελευθερία διέπνε αυτούς τους λαούς ε, και χαίρομαι που οι βασικές πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σε συνενετική λύση και θέλουν να αναδείξουν την Αραβική Άνοιξη ε, και κάποιους από τους πρωταγωνιστές της ε, σε βασικούς πρωταγωνιστές της πολιτικής ζωής. Μοχάμιν Ανσαζή, ένας νέος άσμα μαφούς,

Ε, μία νέα Αιγύπτια, ο ε, Αλή Φαρζάτ ε, από την Συρία και ο Ζαρσάτ Σατουνέ που ενεργοποιούνται στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ο Αχμέτ Ζουμπέρ από τους διάσημους αντιφρονούντες του στρατηγού Γκαντάφη που πέρασε 30 χρόνια στη φυλακή. Όμως πρόκειται για συλλογική δουλειά. Κανένα πολιτικό κόμμα, καμία οργάνωση, καμία ηγετική φυσιογνωμία δεν υπέδειξε την οδό ανατροπή αυτών των απολυταρχικών καθεστώτων. Όλοι έβαλαν το λιθαράκι τους ε, για να οικοδομήσουν την αλλαγή βάσει των ε, ιδιωτήτων τους ε, και βάσει των ικανοτήτων που είχαν. Έτσι δραστηριοποιήθηκαν ε, επιτέλους ε, οι λαοί που είχαν παγώσει εδώ επί σειρά δεκαετιών σε όλες τις χώρες. Ε, τώρα γεύονται όλη την αποκτηθήσα ελευθερία και φυσικά θέλουν να την εγκαταλείψουν. Οι αραβικοί λαοί κατέδειξαν ότι δεν φοβούνται πλέον και δεν δέχονται πλέον την τυφλή εμπιστοσύνη σε απαξιωμένα καθεστώτα. Αγαπητοί συνάδελφοι, να ένα αρκτήριο λάκτισμα, ένα ένασμα. Ο πρώτος νερός ε, την Ίσιος ε, νομίζω ενσαρκώνει αυτή τη νέα πνοή μέσα στον αραβικό κόσμο και γι' αυτό η πολιτική μας ομάδα αποφάσισε ε, να εισηγηθεί την υποψηφιότητά του γιατί συμβολίζει τις ανατροπές που όλοι ζούμε. Ο Μποαζιζή, νέος πτυχιούχος που δεν είχε καταφέρει να βρει δουλειά και που εμπορευόταν οποροκυπευτικά. Ταπεινώθηκε από αστυνομικούς που τον εμπόδισαν να ασκήσει αυτή την απλή επαγγελματική δραστηριότητα. Ζήτησε ακρόαση από το δήμαρχο της πόλης του, όμως αρνήθηκε. Ο δήμαρχος την αίτησε και αυτοπυρπολήθηκε από την απόγνωσή του η Ισία και μεγάλο μέρος του αραβικού κόσμου βλέπει στην άτυχη ιστορία αυτού του νέου ε, τη δική του ζωή και ε, βλέπουμε τη νέα πνοή στον αραβικό κόσμο ε, διότι έτσι τροφοδοτούνται οι ελπίδες μας για το μέλλον και πιστεύω πρέπει να τους συνοδεύσουμε τους αραβικούς λαούς στον δρόμο τους προς μια πιο ισότιμη κατανομή του πλούτου. Βλέπουμε στον Παχρέν, στη Συρία και στην Ιεμένη τις τελευταίες εξελίξεις και αν κρίνω από πρέπει κάθε δύναμη που έχουμε να υποστηρίξουμε αυτόν τον αγώνα. Η απονομή του βραβείου Ζαχάροφ στους πρωταγωνιστές της Αραβικής Άνοιξης ε, αποτελεί αναγνώριση των μαρτυρίων και των δεινών αυτών των λαών και φόρο τιμής προς αυτούς που δεν δίστασαν να θυσιάσουν τη ζωή τους για να καταστήσουν δυνατές ε, αυτές τις αλλαγές. Ε, με αυτές τις μεταρρυθμίσεις μαθαίνουμε ότι χρειάζεται σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ελευθερία της δημοκρατίας είναι κάτι που επιθυμούν οι εταιροί μας από άλλη πλευρά της Μεσογείου ε, οι αρχές αυτές ε, ούτως ή άλλως είναι γεγραμμένο στο DNA μας ε, και άρα θα πρέπει να υποστηρίξουμε αυτούς τους λαούς και θα ήθελα να υποστηρίξετε αυτές τις συμβολικές υποψηφιότητες για την Αραβική Άνοιξη. Ευχαριστούμε κυρία Σαΐφη, η κυρία Βερονίκα Ντεκάιζερ επίσης για τις ίδιες υποψηφιότητες. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα πριν σας μιλήσω για την Αραβική Άνοιξη να πω κάποια λόγια ε, πλέκοντας τα εγκόμια του ε, ε, κυρίου Αμπουλαΐς. Θεωρώ ότι αποτυπώνει το πνεύμα του βραβείου Ζαχάροφ αυτή η υποψηφιότητα φέτος. Ε, επιμείναμε ε, στην, συνενετική, στην εξέβρεση συνενετικής λύσης ανάμεσα σε όλες τις πολιτικές ομάδες για να υπερβούμε ε, τις πολιτικές διχογνωμίες. Όταν ήμουνα στη Γάζα συνάντησα τον κύριο Αμπουλαής, τον έφερα στο Κοινοβούλιο και η συνάντησή του με τον κύριο Πέτερινγκ ήταν από τις πιο συγκινητικές συνθήκες ε, που έχω ζήσει εγώ. Ήδη είχε, είχαμε προτείνει την υποψηφιότητά του πριν από ένα ή δύο χρόνια. Ε, δεν πήρε, ε, δεν κατέλαβε την πρώτη θέση τελικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν πολύ κρωτή η δυο χρονια δεν πηρε δεν καταλαβε την πρωτη θεση τελικα αλλα σε καθε περιπτωση ηταν πολυ κροτή η υποψηφιοτητα του και έλαβε πολλές τιμές κυρίως στη ΣΥΠΑ. Τώρα έχουμε άλλους αγωνιστές της δημοκρατίας και σε αυτούς θα προτιμούσε η πολιτική μου ομάδα ε, να αποδώσουμε μεγαλύτερη σημασία όλοι αυτοί που ε, αγωνίστηκαν για την ελευθερία και τη δημοκρατία στην Αραβική Άνοιξη. Ε, η κυρία Σαϊφά το είπε, πρόκειται για ένα σύμβολο επί της ουσίας, πέρα από τους υποψηφίους, ανθρώπους που είναι αξιόλογοι, όπως και πάρα πολλοί άλλοι ε, πρόκειται όμως για ένα σύμβολο, το σύμβολο της Αραβικής Άνοιξης, του αγώνα για τη δημοκρατία, γιατί επί σειρά δεκαετιών του το αρνούμασταν. Ε, λέγαμε ότι δεν είναι φτιαγμένοι για τη δημοκρατία, μα δεν ισχύει αυτό. Η πολιτική μας ομάδα ε, επέλεξε μία Σύρια πιο συγκεκριμένα για την φετινή υποψηφιότητα που ζει παράνομα στην παρανομία σήμερα η Χαζάν Ζαϊτουνέ ε, και εδώ υπάρχει, υπάρχουν δύο συμβολικές διαστάσεις. Η Συρία ακόμη δεν κατέκτησε την ελευθερία και τη δημοκρατία ε, και είναι ε, αβάστακτη η κατάσταση. Η κυρία Ζέιτουνε φυσικά δεν αγωνίζεται από χθε. Είναι νέα, είναι πάρα πολύ νέα, είναι 34 και πριν από 10 χρόνια ήταν στο κίνημα της Δαμάσε που κατέστηλε το καθεστώς ε, είχε συνεργαστεί με τον Ελμελέ για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συνεχίζει τον αγώνα της στην παρανομία, ξαναλέω. Επλήγει σοβαρότατα διότι ο, ε, συνελήφθη ο άντρα της ε, για, και η και τη ε, για να την εκφοβήσουν. Ε, θα θέλαμε λοιπόν να προτείνουμε την υποψηφιότητα αυτή τη Συρία ε, που δεν υποκύπτει σε καμία πίεση, ακόμη και όταν την πιέζουν μέσω μελών της οικογένειάς της. Υπάρχει και ο περίφημος Αλή Φαρτζά, ε, που που του έσπασαν ε, τα χέρια. Ε, βλέπετε λοιπόν ε, την ομή βία που υπέστη. Συρία λοιπόν, την Ισία αλλά και Λιβύη Έχουμε ολόκληρο το φάσμα της ε, Αραβικής Άνοιξη. βεβαίω έχουμε και την Ιεμένη ε, και τον Μπαχρέιν. Ε, πρόκειται για, ένα, για μια άλλη γεωγραφική ομάδα, αν θέλετε, και ούτως ή άλλως θα ακολουθήσουν και άλλες τιμέ στο μέλλον. Ευχαριστούμε, κυρία Ντεκέζερ. Ευχαριστούμε, Και τώρα, επειδή έχουμε δύο ακόμα τέσσερα από την ίδια πολιτική ομάδα και θα μοιραστούν το χρόνο του. ο κύριο Βάγγελ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η πρόταση να δώσουμε το βραβείο σε πέντε άτομα που συνεισέφεραν στην ε, πρόσφατη επανάσταση, την Αραβική Άνοιξη, είναι αναγνώριση σε όλους τους ανθρώπους που διαδραμάτισαν κάποιο ρόλο. Φοιτητές, ε, bloggers, ε, ακαδημαϊκούς, αγρότες, εργαζόμενους, ε, επικεφαλής αλλά και ε, μέλη της αντιπολίτευσης. Γράφτηκε ένα νέο κεφάλαιο στην ευρύτερη γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, οι άνθρωποι στις αραβικές πόλεις μας βοήθησαν να αναγνωρίσουμε ότι τα στερεότυπα βάσει των οποίων οι Άραβες ε, δεν είναι φτιαγμένοι για τη δημοκρατία και τις σύγχρονες αξίες είναι λανθασμένα. Πρόκειται για στερεότυπα τα οποία αποτέλεσαν απλώς ε, μέσω χειραγώγησης ε, για να διατηρήσουν τη δικτατορία και να διασφαλίζουν μία επίφαση σταθερότητας της περιοχής. Οι νέοι Άραβες προσέγγισαν τον κόσμο. Πρόκειται για νέους ε, τους οποίους εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν μπορούσαμε να κατανοήσουμε και μας απέδειξαν ότι οι κοινέ αξίες μεταξύ των οποίων η ελευθερία και η δημοκρατία, ο σεβασμός ε, της ιδιαιτερότητας ε, του καθενός, των γυναικών, των παιδιών, των μειονοτήτων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εν γέννη, είναι κάτι για το οποίο πρέπει να είμαστε έτοιμοι να θυσιαστούμε, να θυσιάσουμε ακόμα και τη ζωή μας. Η Αραβική Άνοιξη αποτελεί με ένα ψήγμα ελπίδας ε, και μια δημιουργικού και ειρηνικού γειτονικού κόσμου σε εμά. Ευχαριστώ και τώρα η κυρία Σάκη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο πάρα πολύ θα συμφωνήσω και εγώ με τους προλαλήσαντες ε, συναδέλφους και θα ήθελα να τονίσω την Ασμά μαχφουζή Είναι ένα από τα σύμβολα που εκπροσωπεί τους ε, πολλούς ανθρώπους στην ε, Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή και είχα την ευκαιρία να συναντήσω πολλούς από αυτούς τους τελευταίους μήνες στην Αίγυπτο, πολλούς ακτιβιστές, για να κάνω και εγώ έτσι λίγο μια εκστρατεία και να μοιραστώ κοινοβουλευτική εμπειρία. Είναι μια νεαρή φοιτήτρια, 26 ετών, ξεκίνησε να χρησιμοποιεί το YouTube και ε, Βεβαίω ανέβασε δύο βιντεοκλίπ τα οποία αποδείχθηκαν πάρα πολύ επίκαιρα και επηρέασαν πάρα πολύ. Εκεί πέρα μιλούσε για την δικαιοσύνη, την ελευθερία και τα ίσα δικαιώματα και καλούσε ιδιαίτερα τις γυναίκες να ε, συνταχθούν μαζί της. Μαζί με πάρα πολλά άτομα που ε, ψήφισαν τον φόβο, πήγαν στην Ταχριέρη στις 26 Ιανουαρίου και τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Αυτή η γυναίκα εκπροσωπεί τη νέα γενιά μιας διαφορετικής Αιγύπτου. Είναι το μέλλον αβέβαιο, βεβαίω, αλλά ακτιβιστές ε, σαν και εκείνοι, με το θάρρος της γνώμης τους, ε, επικριτικοί, είναι πάρα πολλοί και καθορίζουν μαζί το μέλλον της χώρας τους, το οποίο δεν θα είναι εύκολα, αλλά θα έχει αυτούς τους νέους ηγέτες. Ε, το ότι μιλάει ανοιχτά της, έχει βεβαίως δημιουργήσει νέους φίλους, αλλά και πάρα πολλούς επικριτές και την ε, ανέκρινε το Ανώτατο Συμβούλιο των Ανόπλων Δυνάμεων, το οποίο αυτή τη στιγμή ασκεί την εξουσία στην Αίγυπτο. Αφέθηκε ελεύθερη και έχει συνεχίσει την εκστρατεία ε, για να σταματήσουν να δικάζονται οι πολίτες σε στρατιωτικά δικαστήρια, την οποία ξέρω πως πολλοί εδώ μέσα υποστηρίζουν. Εν ολίγης, αυτή η νεαρή γυναίκα εκπροσωπεί τη νέα γενιά της Αιγύπτου που αψήφισε τον φόβο και ζήτησε ίσα δικαιώματα, αυτοδιάθεση, ευκαιρίες και ελευθερίες. Η χρήση βεβαίως των νέων αυτών μέσων είναι μέρος της υποσφιότητάς της και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή η ελευθερία σκέψης και η ελευθερία έκφρασης ε, σχετίζονται. Είναι ένα σημαντικό σύμβολο μαζί με τους υπόλοιπους ε, σεβαστούς υποσφίους ε, που καλούμε συλλογικά Αραβική Άνοιξη και ελπίζω να βρει στήριξη διακομματική εντός του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Ελέν Φλότρα. Ελέν Φλότρα έχει το λόγο. Merci, Madame la Présidente. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, προφανέστατα δεν ε, εκπλήσεται κανείς που Θέλουν οι συνάδελφοι να ρίξουν τα φώτα της δημοσιότητας ε, στους πρωταγωνιστές των αραβικών ε, επαναστάσεων ε, για να προβάλλουν την ελευθερία έκφρασης, την ελευθερία συνείδησης που είναι στον πυρήνα του βραβείου Ζαχάροφ. Πονέμοντας το βραβείο στους πρωταγωνιστές αυτής της δράσης πρόκειται για ένα συλλογικό έργο. Το αποτέλεσμα φυσικά ήταν απελευθέρωση αυτών των λαών. Είναι ενδιαφέρον να τονίσουμε το ότι η ελευθερία έκφρασης παρήγαγε ένα, μια απίστευτη ενέργεια σε αυτούς τους λαούς η οποία μεταδόθηκε ε, ε, μέσα από ένα κύμα σε άλλες χώρες και μέσα από αυτό το κύμα και τα κοινωνικά δίκτυα επικοινωνούν πλέον αυτές οι χώρες. Θα ήθελα να τονίσω επίσης ότι όταν η καταστολή των επαναστάσεων όπως αυτό που ζούμε σήμερα στη Συρία ε, όταν γίνεται αυτή λοιπόν η καταστολή και κλεισμένων ε, των θύρων ε, με στόχο την φυλάκιση, την απαγόρευση της επικοινωνίας με τον έξω κόσμο, λοιπόν οι δράσεις που αναλαμβάνονται όπως αυτή την στο σελίδα του Χαζάς Ουζετινέ στην Συρία για να έχουμε τις ακριβέστερες δυνατές πληροφορίες για όσους έχουν φυλακιστεί κτλ. Λοιπόν, πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο και το τον αποντάρουμε ε, όπως ε, το έκανε στην ενημέρωση, στην κυκλοφορία των πληροφοριών ε, και τη χρήση των πληροφοριών ως κινητήριο δύναμη της Επανάστασης. Είναι μια εκπληκτική ιδέα το βραβείο Ζαχάροφ δεν ε, ε, αποτελεί απονομή έτσι, μιας αμοιβή, ε, δεν ενθρονίζουμε κανέναν, υποστηρίζουμε τους υπερασπιστές των δικαιωμάτων που στη Συρία και σε άλλες χώρες ρηψοκινδυνεύουν τη ζωή τους για να αγωνιστούν κατά της καταστολής με τρόπο ώστε η διεθνής κοινότητα να δραστηριοποιηθεί. Πρέπει να είμαστε στο ύψος των επιθυμιών και των φιλοδοξιών αυτών των ανθρώπων. Ε, ξέρετε, δεν έχει ολοκληρωθεί η Αραβική Άνοιξη. Ε, το κύμα δεν έχει φτάσει ακόμη στην Ευρώπη και στους, στα δικά μας ε, θεσμικά όργανα. Ε, δεν έχουμε διαβάσει το τέλος της ιστορίας. Ας σταθούμε λοιπόν στο ύψος των φιλοδοξιών τους και το βραβείο Ζαχαρόφ αν τιμήσει τους πρωταγωνιστές της Αραβικής Άνοιξης ε, θα μας δείξει ότι αναγνωρίζουμε την αξιοπρέπειά τους, ε, το έργο τους ε, και ποντάρουμε σε αυτούς, δηλαδή τους εμπιστευόμαστε ουσιαστικά για τον τρόπο με τον οποίο θα επινοήσουν τη νέα οδό προς τη δημοκρατία, προς την ανάπτυξη και θα ήθελα να επιμείνω σε αυτό διότι ξαναλέω ότι μπορεί να έχουμε αυτά τα πολύ άσχημα και αντιδραστικά αντανακλαστικά, προκάτε ε, αντανακλαστικά που θα επιβληθούν τελικά από εμά. Περιμένουν να τους ακούσουμε, να τους ε, δείξουμε εμπιστοσύνη, να έχουμε ανοιχτό μυαλό. Και λοιπόν, ε, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να περάσουμε αυτό το μήνυμα στους πρωταγωνιστές της Αραβικής Άνοιξης ευχαριστώντας τους για αυτό που ήδη έχουν καταφέρει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η τελευταία παρουσίαση είναι από την κυρία Πράντινα. Ναι, ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Έγιναν πολλά σχόλια για την κοινή προσέγγιση που αποτελεί αφενός εορτασμό και ταυτόχρονα ενθάρρυνση των όσων συνέβησαν ε, στην Αφρική όλοι ενθαρρύνουν ε, το δικαίωμα για την ελευθερία του λόγου και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών αυτών των χωρών. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι είναι μια διαδικασία εν εξελίξη. Δεν μπορούμε να πούμε σε καμία από τις χώρες ότι τελειώσαμε, μπορούμε να γυρίσουμε σπίτια μας, ε, τελείωσαν όλα. Πολλέ από αυτέ τι χώρε βρίσκονται ακόμα σε πονίδιστε συνθήκε, όπω για παράδειγμα η Συρία, αλλά και άλλε και επομένως το βραβείο αυτό θα αποτελέσει και ένδειξη υποστήριξης και ταυτόχρονα και επίκρισης ε, προς όλες αυτές τις δυνάμεις που προσπαθούν να σταματήσουν ε, τα κινήματα αυτά και ε, να μην τα αφήσουν να οδεύσουν εκεί που πρέπει να οδεύσουν. Άκουσα και από άλλους ευρωπαϊκούς φορούς ε, ε, επικρίσεις για το πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Ε, εμείς πρέπει να δώσουμε ένα μήνυμα πολυφωνίας. Ε, οι νέοι άνδρες και γυναίκες ε, πρέπει να συνεχίσουν ε, να, το έργο τους και το πιο σημαντικό είναι να επιστρέψουμε στη σταθερότητα και εμείς να συνεχίσουμε να τους πιστεύουμε. Ακούσαμε λοιπόν όλες τις παρουσιάσεις τώρα οι οποίες σχετίζονται με την κοινή υποψηφιότητα της Αραβικής Άνοιξης και τώρα περνάμε στην επόμενη ο κύριος Μικάλσκι έχει το λόγο και νομίζω ότι θέλετε να δείξετε και ένα βίντεο. Ελπίζω λοιπόν να είναι έτοιμο το βίντεο σας. Κύριε Μικάλσκι. Καλημέρα κυρίες μου και κύριοι. Έχω τη μεγάλη τιμή να σας παρουσιάσω εδώ πέρα τον Δημήτρη Μπανταρένκα αντιπολίτευση, μέλος της αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία αυτή τη στιγμή είναι φυλακισμένος έχει καταδικαστεί σε δύο χρόνια φυλάκιση βλέπετε εδώ πέρα διαδήλωση μετά την 19η Δεκεμβρίου 2010 μετά τις προεδρικές εκλογές όταν συνελήφθησαν εκατοντάδες άνθρωποι στη Λευκορωσία και συνελήφθησαν όλοι οι ανθυποψήφοι του Λουκασέγκο. Πράγματα ανήκουστα. Μεταξύ άλλων συνελήφθηκε ο κύριος Δημήτρη Μπανταρενκό που ήταν επικεφαλής του εκλογικού επιτελείου ενός ανθυποψηφίου. Είναι δραματική η κατάστασή του στη φυλακή αναγκάστηκε να υποστεί εγχείρηση στην σπονδυλική του στήλη χωρίς μέτρα ανάνυψης και αποκατάστασης και μετά τον έστειλαν απλά σε ένα στρατόπεδο και η γυναίκα του ε, αναγκάστηκε να κάνει καθιστική διαμαρτυρία μπροστά από ένα κτίριο δημόσιο για να μην μεταφερθεί στο στρατόπεδο σύζυγός της για να όπου δεν θα μπορούσε να κάνει βεβαίως καμία αποκατάσταση και κινδυνεύει η ζωή του. Οπότε αυτό το βραβείο, αυτή η υποψηφιότητα μπορεί να σώσει τη ζωή αυτού του ανθρώπου. Δεν είναι μόνο ένα μήνυμα που θα στείλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον Λουκασέγκο. Μιλάμε για τον τελευταίο παραδοσιακό δικτάτορα στην Ευρώπη άνθρωπο που δολοφονεί, πολεμά την αντιπολίτευση, δεν ανέχεται καμία ελευθερία. Πρέπει να δείξουμε πως δεν δεχόμαστε τέτοια πράγματα στη γειτονιά της Ευρώπης. Η Λευκορωσία είναι γείτονάς μας. Εάν δεν αντιδράσουμε θα εξευτελιστούμε. Αντιθέτως ο Λουκασέγκο θα ενθαρρυνθεί να κάνει ό,τι θέλει. Ο κύριος Μπανταρένκα ε, συμμετέχει στην αντιπολίτευση εδώ και χρόνια, ίδρυσε ένα πόρταλ, το Χάρτα 76 και, και ο webmaster ε, της σελίδας αυτής επίσης εξαφανίστηκε και δεν ξέρουμε τι του συνέβη. Η, σύζυγάς, η σύζυγός του, η Όλγα Μπανταρέκα, Επίσης ε, συμμετέχει σε ένα κίνημα των ε, οικογενειών των ε, συλληφθέντων όπως και η κόρη του συμμετέχει σε αντιπολιτευτικές δραστηριότητες. Ολόκληρη η αντιπολίτευση στην Λευκορωσία προσπαθεί να παλέψει για την απελευθέρωση των συλληφθέντων. Αυτό είναι το βασικό, ο βασικότερος στόχος της αντιπολιτευσής. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για τον Μπανταρένκα Μπορούμε να τον στηρίξουμε με τον τρόπο αυτό και θεωρώ πως αν λάβει το βραβείο Ζαχάροφ θα αποτελέσει αυτό ισχυρό μήνυμα και θα έχουμε δύο διαστάσεις πρώτα απ' όλα συγκεκριμένη βοήθεια προς τον κύριο Μπαναρέγκο του οποίου η ζωή κινδυνεύει όπως σας είπα και δεύτερον είναι ένα μήνυμα το, των αξιών τις οποίες ε, υπερασπιζόμαστε ότι δεν θα δεχτούμε οι δικτάτορες να κάνουν ό,τι θέλουν στην χώρα τους. Θα δείξουμε πως είναι σημαντικό για εμάς ε, ε, και η Λευκορωσία να μοιράζεται τις ευρωπαϊκές αξίες. Και τέλος, θα πω το εξή, όποιο σώζει μια ζωή σώζει τον κόσμο όλο. Και εδώ πέρα έχουμε τη δυνατότητα να σώσουμε μια ζωή και ταυτόχρονα μπορούμε να σώσουμε την τιμή μας και την ε, αίσθηση πως είμαστε αξιοπρεπείς. Πως είμαστε σε θέση όχι μόνο να έχουμε πολιτικούς στόχους αλλά και ανθρωπιστικούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Yes. Thank Ευχαριστώ αγαπητοί πρόεδροι των Επιτροπών, αγαπητοί συνάδελφοι. Με θυμάται ότι έχω σήμερα τη δυνατότητα να παρουσιάσω μία από τις πέντε υποψηφιότητες για το βραβείο Ζαχάροφ, τον κύριο Μπόρις Παχόρ. Ο Παχόρ έλαβε υπογραφές ε, και στήριξη από 52 μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από 17 χώρες μεταξύ των οποίων 9 επικεφαλής αντιπροσωπιών. Θεωρούμε λοιπόν άρα πως έχουμε μια πολύ ισχυρή υποψηφιότητα. Ο κύριος Μπόρις Πάχορ είναι συγγραφέας, αγωνίζεται για την ελευθερία σκέψης, ε, υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ε, θεμελιώδεις ελευθερίες, ε, υπερασπίζεται τις μειονοτικές γλώσσες και τα δικαιώματα των μειονοτήτων, είναι ακέραιος και γεννήθηκε το 1900 1930. Είναι Σλοβαίνος ε, και έχει και σλοβενική και Ιταλική υπηκοότητα. Θεωρείται πως είναι ένας από τους πιο σημαντικούς ε, Σλοβαίνους συγγραφείς στην ζωή. Έχει γράψει στα Σλοβενικά, στα Ιταλικά και στα Γαλλικά και έχει λάβει πολλά βραβεία. Λογοτεχνικά και η συνεισφορά του μεταξύ άλλων ε, έχει οδηγήσει στο να χρηστεί υπό της, ε, της λεγεώνας της τιμής από την γαλλική κυβέρνηση. Μεταξύ άλλων ε, παρασύμων, επίσης ε, σταυρός πρώτης τάξεως στο τάγμα των γραμμάτων και των τεχνών από την Αυστρία και επίσης έχει παρασημοφορηθεί από την Γερμανία και ήταν υποψήφιος για το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Επίσης ε, επέζησε από στρατόπεδο συγκέντρωσης και πάντα ήταν αντίθετο στον φασισμό. Η εμπειρία του στο στρατόπεδο συγκέντρωσης ε, απετέλεσε μεγάλη έμπνευση και το λογοτεχνικό του έργο βεβαίω ε, συνδέεται στενά με την εμπειρία του για με την του πρώτου μισού του παγκοσμίου του 20ου αιώνα, Επίσης, ήταν πάντα κατά του κομμουνιστικού καθεστώτος της Ιουγκοσλαβίας, ίδρυσε ένα περιοδικό στο οποίο έγραφε τις ε, απόψεις του. Επίσης, ο Γάλλος πρεσβευτής στη Σλοβενία δήλωσε γι' αυτόν «Η ζωή σας ε, έχει σημαδευτεί από το θάρρος και την επιμονή σας να παλεύετε ενάντια σε κάθε μορφή απολυταρχίας και όμως η φιλοσοφία σας ονομάζεται ανθρωπισμός. Η πρέσβης εξέφρασε την ε, πεποίθησή της πως η Νεκρόπολης ε, που γράφηκε το 67 και μεταφράστηκε στα γαλλικά το 1990 αποτελεί την ε, πιο συγκινητική μαρτυρία της ναζιστικής θηριωδίας. They Κυρίε και κύριοι, όλοι οι φετινοί υποψήφοι είναι βεβαίω αξιοί να κερδίσουν το βραβείο. Τα μέλη της ε, σλοβενικής αντιπροσωπείας ε, στο ΕΛΚ, ε, Γιώργαν Σίσιλ και Πέτερ Λέντα, χαίρονται για το ότι έχουν συμπατριώτη αυτόν τον άνθρωπο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ευχαριστούμε κύριε Τσβέρ. Ο Κλούτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια που η συνάδελφος η Μαρία Κριστίν Βερζιά απουσιάζει θα παρουσιάσω εγώ την υποψηφιότητά μας για το βραβείο Ζαχάροφ. Το βραβείο Ζαχάροφ θα πρέπει να τιμά ανθρώπους οι οποίοι μάχονται για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Και βεβαίως ε, επειδή ο αγώνας αυτός είναι πάντα δύσκολος, το βραβείο αυτό παίζει και ένα ρόλο προστασίας αυτών των ανθρώπων. Για να μπορέσουμε λοιπόν καλύτερα να παρουσιάσουμε το φετινό μας υποψήφιο θα σας δείξουμε κάποιες εικόνες. Αλλά γιατί ε, κάποιον από την Πολωνία. Η Πολωνία είναι μια πολύ πλούσια χώρα στην Νότια Αμερική αλλά ταυτόχρονα ζει μια μεγάλη τραγωδία εδώ και 16 χρόνια μένεται ένας εμφύλιος ε, πόλεμος ε, στον οποίο σκοτώνται αυτό οι πολίτες της χώρας. Το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο απαιτεί από τους ε, εμπολέμους να σεβαστούν τους άμαχους και να κατευθύνουν επιχειρήσεις μόνο εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Παρόλα αυτά ο πόλεμος διεξάγεται κυρίως εις βάρος των αμάχων στην ε, Κολομβία και μάλιστα ιδιαίτερα εις βάρος των μικροαγροτών. Έχουμε γύρω στους 38 ε, εξαφανισμένους, γύρω ανθρώπους τα τελευταία τρία χρόνια. Μιλάμε για πάνω από 3 εκατομμύρια εσωτερικούς προσφύγους, ε, αριθμοί πολύ χειρότεροι από πολλές δικτατορίες της ε, Λατινικής ε, Αμερικής. Οπότε προτείνουμε το Σαν Χωσέ Δε Απαρτάδο για το βραβείο Ζαχάροφ του 2011. Πρόκειται για μια κοινότητα στην οποία οι μικροκαλλιεργητές, οι καμπεσίνος αποφάσισαν να ζήσουν ειρηνικά και να μην εμπλακούν με καμία πλευρά της ε, σύγκρουσης. Μιλάμε για μικροκαλλιεργητές που είχαν την ε, ατυχία να βρίσκονται κοντά στα σύνορα με τον ε, Παναμά. Οπότε πηγαίνουν τα ναρκωτικά προς βοράν και τα όπλα προς νότον. Ούτως ή υπήρχε βία από το 1980 και είδαν πως το κράτος δεν μπορεί να τους προστατεύσει οι υπόλοιπες ε, γεωργικές ε, κοινότητες ε, αναγκάστηκαν να μπουν σε κάποια από τις δύο πλευρές του εμβυλίου. Αντιθέτως παρέμεινε ουδέτερο αυτό το χωριό, απαγορεύονται αυστηρά τα όπλα, δεν υποστηρίζει ούτε αντάρτες ούτε παραστρατιωτικούς, παρόλα αυτά έχουν χάσει πάνω από 180 ανθρώπους τα τελευταία χρόνια στο χωριό αυτό. Η, τιμή, η τιμή στους ε, νεκρούς αυτούς ε, και στο χωριό αυτό θα αποτελέσει σημαντικό κομμάτι και ένδειξη αλληλεγγύης. Εμείς λένε αυτοί οι άνθρωποι πως εμείς δεν απαιτούμε καμία εκδίκηση, θεωρούμε πως κάθε βία είναι πόλεμος και έχουμε κάνει αυτή την επιλογή για το χωριό μας. Ε, καθημερινότητά τους χαρακτηρίζεται από απειλές ε, θανάτου αλλά και προσπαθούν, όπως είπαμε, να μεταδώσουν αυτές τις αξίες στα παιδιά τους. Ε, επίσης υπάρχει και ένα σχετικό σχολείο, ένα πανεπιστήμιο θα λέγαμε που διοργανώνεται εκεί πέρα, το οποίο στηρίζεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά το ότι λοιπόν η σύγκρουση στην Κολομβία συνεχίζεται, τα μέλη του στρατού και παραστρατιωτικοί το 2005 προέβησαν σε σφαγές ε, στο Σαν και κατέληξαν στο να δικαστούν η ομάδα μας ε, θεωρεί πως ε, χρειάζονται τέτοιοι άνθρωποι στην Κολομβία για να βρεθεί μια διέξοδος από την βία. Η, αναξόριση από το, η αναγνώριση από το εξωτερικό είναι κάτι σημαντικό και μπορεί να δώσει όθηση. Όπως ξέρετε έχουν ήδη εγκατασταθεί πέντε παραστρατιωτικές ομάδες στο έδαφος ε, της κοινότητάς τους και κάποιοι άνθρωποι από αυτό το χωριό έχουν έρθει στις Βρυξέλλες και θα είναι στην διάθεσή σας για ερωτήσεις και για να σας ευχαριστήσουν για την υποψηφιότητα αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κλούτε και νομίζω ότι τώρα ακούσαμε πάρα πολύ καλές και εντυπωσιακέ παρουσιάσεις, διαφορετικές μεταξύ τους, αλλά είναι εξέχουσες όλες αυτές οι φυσιογνωμίες που περιγράψατε. Θα ήθελα να Δώσω τώρα το, την Προεδρία στην ε, κυρία Κρετή που εκπροσωπεί την Επιτροπή Ανάπτυξης ε, για να ακολουθήσει μια σύντομη συζήτηση για το θέμα. Ε, μισή ώρα έχουμε στη διάθεσή μας για να κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση για όλους όσους είχαν κάτι να σχολιάσουν. We have the πριν ε, ακούσουμε τα συμπεράσματα της ε, συζήτησης. Θα ήθελε κάποιος το λόγο παρακαλώ. So I think we... Uh, Μάλιστα. Αν ε, δεν γίνει συζήτηση, Μπορώ να σας ε, ευχαριστήσω όλους που υποστηρίξατε τους υποψηφίους σας. Ε, φυσικά είναι όλοι πολύ καλοί υποψήφοι, αλλά θα πρέπει να βρούμε την ευρύτερη δυνατή συνένεση για τον υποψήφιο ως γνωστόν. Θα μπορούσαμε να μείνουμε εδώ μέρες ε, και μήνες ε, για να μιλάμε για άντρες ε, και γυναίκες που αγωνίζονται για την ελευθερία αλλά το βραβείο Ζαχάροφ είναι για την ελευθερία του λόγου, την ελευθερία συνείδησης όποιος και αν επιλεγεί Είμαι σίγουρη ότι ο υποψήφιος θα ενσαρκώνει το πνεύμα του βραβείου Ζαχάροφ που έχει η οικονομία το οποίο ξεκίνησε το 1988. Στις 4.30 θα μας επισκεφθεί ο Γενικός Διευθυντής της UNICEF, ο κ. Άντωνη Λέικ, αλλά πριν κλείσουμε ε, τη συνεδρία θα σας υπενθυμίσω το χρονοδιάγραμμα. Ε, για, τον, ε, ε, για τους τρεις υποψηφίους την 5η στις 30 Οκτωβρίου το πρωί στην Κοινή Επιτροπή στην Κοινή Συνεδρία των Επιτροπών θα γίνει η πρώτη ψηφοφορία μετά στις 27 Οκτωβρίου στην, στο Στρασβούργο θα γίνει η ψηφοφορία και στις 12 Δεκεμβρίου τη Δευτέρα στο Στρασβούργο θα καλέσουμε τους υποψηφίους ε, και την Τετάρτη στις 14 Σεπτεμβρίου στις 12 στο Στρασβούργο θα γίνει η τελετή απονομής και ε, θα ε, μεριμνήσει η Γενική Γραμματεία του ε, Κοινοβουλίου για την προβολή της τελετής. Θα υπάρχουν εκδηλώσεις όχι μόνο στο Κοινοβούλιο, μέσα και έξω, αλλά και στην πόλη. Ευχαριστώ και στις 4.30 θα συνεχίσουμε με τον Γενικό Διευθυντή της UNICEF.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

Ευχαριστώ.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

Um, ε, νομίζω πως πρέπει να ξεκινήσουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, με ιδιαίτερη ευχαρίστηση σήμερα καλωσορίζω τον εκτελεστικό διευθυντή της UNICEF, τον Άντωνη Λέι, και έχουμε την τιμή να τον έχουμε εδώ για μια ανταλλαγή απόψεων σε μια κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Ανάπτυξης και την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Καλωσορίζω λοιπόν τα μέλη που είναι παρόντα από αμφότερες επιτροπές. Ο Διευθυντής Αντωνι Λέικ δεν χρειάζεται συστάσεις. Στα 45 χρόνια δημόσιου βίου συνεργάστηκε με επικεφαλής ε, ε, αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων από όλο τον κόσμο. Ήταν ε, υπεύθυνος της προεκλογικής εκστρατείας ε, με την ε, ε, επακόλουθηση επιτυχία του Πρόεδρου Ομπάμα. Ήταν συνεργάτης επίσης του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον και στη σταδιοδρομία του ασχολήθηκε με πολύ περίπλοκα πράγματα, ιδίως όσον αφορά ανθρωπιστικά και αναπτυξιακά ζητήματα. Οι σχέσεις του με τη UNICEF χρονολογούνται από πολύ παλιά και ε, ανέλαβε καθήκοντα διευθυντή από τον περασμένο Μάιο. Με την ε, συνθήκη της Λισαβόνας, να κάνω μια σύντομη εισαγωγή στο θέμα που θα μας αναπτύξετε, η μέρημνα για τα δικαιώματα των ανηλίκων είναι ένα από τα εγκάρσια ε, θέματα αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα πρέπει να το προωθήσουμε τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική του διάσταση. Θέλουμε λοιπόν να προάγουμε και να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των παιδιών και αυτό έχει γίνει ένα απόσπαστο τμήμα της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και φυσικά θα πρέπει να το παραπέμψουμε και στις πτυχές που σχετίζονται με την ασφάλεια, την ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Από πλευράς ασφάλειας οι προκλήσεις για τη ζωή των παιδιών είναι πολλαπλές. Ε, πολλές φορές υπάρχει η φρικτή συμμετοχή τους σε ένοπλες σειράξεις, η χρήση των παιδιών ως εργατικό δυναμικό χαμηλού ε, κόστους, ε, ε, τα παιδιά στρατιώτες, ε, σεξουαλικά κλίματα κατά των παιδιών σε ένοπλες σειράξεις, παιδιά τα οποία έχουν σχέση με ένοπλες ομάδες και στρατιωτικές ομάδες. Ε, και αυτό ε, είναι κάτι το οποίο μας οδηγεί στο να λάβουμε μέτρα και να δώσουμε αποτελεσματικές απαντήσεις ε, για τα όσα ζουν τα παιδιά και σε τι συνθήκες βιώνουν και χαιρόμαστε που θα σας ακούσουμε διότι ε, θα μας δώσετε και κάποιες προτάσεις για το πώς η διεθνή κοινότητα με τη συνδρομή της UNOSIF μπορεί να κάνει τη ζωή των παιδιών καλύτερη. Επειδή δεν είναι πολύ ε, αθρώα η παρουσία των ε, συναδέλφων, ε, αν και βλέπω ότι σιγά σιγά έρχονται, δεν υπάρχει κάποιος χρονικός περιορισμός, σας ακούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ κύριε Αλμπερτίνη. Κυρία Κρέτου, κυρία Λόχμπιλε, Θα είμαι παρόλα αυτά σύντομο σχετικά, παρότι έχουμε τόσα πολλά που μπορούμε να πούμε. Αρχίζοντας, θα ήθελα να τονίσω πόσο εκτιμά η UNICEF την εταιρική σχέση που έχει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χθε είχα επαφές με την ε, Επίτροπο Γεωργίωβε και τον Επίτροπο Πίμπαλξ και εντυπωσιάστηκα από την ποιότητα των επαφών μας. Ε, η προσήλωση Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής για την ανθρωπιστική δράση και την αναπτυξιακή δράση έχει κέρια σημασία για τις διεθνείς προσπάθειες που γίνονται σε αυτό το τομέα. Είναι αυξανόμενο το ενδιαφέρον ε, και προσέβλεπω μια ανυπομονησία στη σημερινή μα συνάντηση. Η εταιρική μας σχέση καθοδηγείται από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών η συνθήκη της Λισαβόνας ενίσχυσε τη σχέση αυτή και επίσης από τη δρομολόγηση της συμμαχία για τα παιδιά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χάρη στην οποία ε, στην καρδιά όλων των πολιτικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βρίσκονται τα παιδιά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η UNICEF έχουν ένα κοινό όραμα για να ενισχύσουν και να σώσουν τη ζωή των ε, απόρων, των παιδιών που το χρειάζονται περισσότερο. Ε, έχουμε, είμαστε προσιλωμένοι, θέλουμε να έχουμε αποτελέσματα γιατί εν τέλει αυτό έχει σημασία ε, στην προσπάθεια που κάνουμε για να προαγάγουμε τα δικαιώματα των παιδιών. Σήμερα θα ήθελα να σας πω πώς η UNICEF και οι εταίροι της εργάζονται για να επιτύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Για να ε, ε, παραφράσω έναν υπέροχο Λιβανέζο ποιητή Χαλίλ Κιμπράν, ναι, η πρόοδος δεν έγκυται τόσο πολύ στην ενίσχυση ε, αυτά, αυτών που ισχύουν, αλλά στην πρόοδο προς αυτά που θα έπρεπε να ισχύουν. Για να επιτύχουμε αυτό το στόχο, θα πρέπει να βρούμε τα παιδιά, ακόμη και όταν είναι δύσκολο, να τα βοηθήσουμε όταν έχουν αναπηρίες, όταν ε, ζουν ε, κρυμμένα, να ε, ενισχύσουμε την δράση των αυτόχθων πληθυσμών για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών, να βοηθήσουμε τα παιδιά που βρίσκονται μέσα σε ένοπλες σειράξεις. Για πολλά χρόνια και ακόμη περισσότερο σήμερα οι ειδικοί στον αναπτυξιακό τομέα θεωρούσαν ότι ήταν υπερβολικό το Κόστο, για να βρούμε ποια είναι τα παιδιά που βρίσκονται στη δυσμενέστερη θέση. Μα έλεγαν ότι θα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα βοηθώντας ε, αυτού που ήταν πιο εύκολο να βοηθήσουμε. Υπήρξαν αποτελέσματα όμω, σημειώθηκε πρόοδο και βοηθήσαμε όντω πολλά παιδιά, αλλά όχι αρκετά και όχι όλα τα παιδιά κυρίως. Ε, η διεθνή ε, κοινότητα αρχίζει να αποτιμά τώρα την πρόοδο προ την επίτευξη των στόχων τη χιλιετία και ανακαλύψαμε ότι η πρόοδος μας ε, ε, μετρημένη με εθνικούς μέσους όρους ε, κρύβει θύλακους, θύλακες απόγνωσης και διευρυνόμενα χάσματα, ανισότητες. Χρησιμοποιούμε τώρα ένα πρότυπο για να αναθεωρήσουμε την κατάσταση διότι βλέπουμε ότι ε, συνειδητοποιούμε ότι υπάρχουν μεγάλες ανάγκες ε, στις ε, λιγότερο ευνοημένες περιοχές, αλλά αναρωτιόμαστε αν κάνουμε αυτές τις προσπάθειες, όμως θα είναι υπερβολικό το κόστος. Θεωρούμε όμως μετά από την ενδελεχή αυτή ανάλυση ότι δεν είναι αυτός ο σωστός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε. Πρέπει να ακολουθήσουμε έναν ευφιέστερο δρόμο, ένα πιο πρακτικό δρόμο για να βοηθήσουμε τα παιδιά. Παραδείγματος χάρη, για χώρες όπου είναι χαμηλά τα εισοδήματα και υψηλή ηθνησιμότητα, ε, ε, κάθε επιπλέον ευρώ ή εκατομμύριο ευρώ που ε, επενδύεται μπορεί να βοηθήσει τα πλέον ευάλωτα παιδιά και μπορεί, αν αλλάξουμε την προσέγγιση μας, να βοηθήσουμε έως και 60% περισσότερα παιδιά και να αποτρέψουμε τους αντίστοιχους θανάτους. Αν ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο θα έχουμε μεγαλύτερα πλέον και μεγαλύτερο αριθμό παιδιών. Μέσα από την οργάνωσή μας η UNICEF να υιοθετεί αυτή τη νέα προσέγγιση που ε, ε, συμβαδίζει με την ατζέντα για αλλαγή. Μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαρτογραφούμε τους το, τις χώρες, τις περιοχές όπου υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες, βγάζουμε νέους μέσους όρους και βλέπουμε πώς θα ε, αγγίξουμε τα παιδιά σε δυσπρόσβατα σημεία ε, προσπαθούμε να λειτουργήσουμε σε διάφορου ε, τομεί και κυρίω να αγγίξουμε χώρε ε, που βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση από πλευρά απόσταση και δημογραφικών χαρακτηριστικών. Επίση, έχουμε αυξήσει τον αριθμό των ανθρώπων που επιτόπου βοηθούν τι οικογένειε και τα παιδιά που το χρειάζονται περισσότερο. Κάνουμε μια καλύτερη αξιολόγηση αποτίμηση των προγραμμάτων μα για να δούμε ποια προγράμματα έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα και να διαπιστώσουμε πού χρειάζονται επιπρόσθετη πόρη Χρειάζεται καλύτερη παρακολούθηση των αποτελεσμάτων για να διαχειριζόμαστε καλύτερα τι προσπάθειε που κάνουμε για να επιτύχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Θα ήθελα λοιπόν να μοιραστώ μαζί σας κάποια παραδείγματα αυτή τη δουλειά που κάνουμε και στην πράξη θα αποδείξουμε πέρα από, από το, αυτά που ισχύουν επί της αρχή ότι η επίτευξη τη ισότητα είναι μονόδρομος. Θα ήθελα λοιπόν ε, να αρχίσω Ε, τη διακοπή της ανάπτυξης ε, των παιδιών ε, λόγω του υποσυτισμού είναι μόνιμες οι βλάβες που προκαλεί. Αυτά τα παιδιά δεν μπορούν ποτέ να μάθουν ή να μάθουν όσα θα μπορούσαν να μάθουν αν είχαν τραφεί σωστά στα πρώτα χρόνια της ζωής τους και ανά τον κόσμο περίπου 175 εκατομμύρια παιδιά πλήττονται σχεδόν εφταπλάσιος αριθμός σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό των παιδιών κάτω των 5 ετών. Και βάσει της συνεδρικής λύσης της Κοπενχάγης οι μικροθρεπτικές ουσίες, ε, βιταμίνη α, ε, ψευδάργυρος, ε, σίδηρος κτλ. Είναι πράγματα που δεν συνεπάγονται μεγάλο κόστος και εύκολα μπορούμε να προμηθέσουμε σε αυτά τα παιδιά και είναι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος για να ενισχύσουμε την παγκόσμια ευημερία. Το 2005 στο Περού, όπου 40% περίπου όλων των παιδιών στην Ήπεθρο υποφέρουν από αυτό, η κυβέρνηση ξεκίνησε ένα επιστημιστικό πρόγραμμα στις ε, φτωχότερες ε, περιοχές ε, τους υπαίθρου και σημειώθηκε μείωση 10%. Χιλιάδες παιδιά μπόρεσαν να παρακολουθήσουν καλύτερα το σχολείο και να ζήσουν καλύτερα, να κερδίσουν τα προστοζήν για την οικογένειά τους και να συμβάλλουν στη συνέχεια στην κοινωνία. Χάρη στην εταιρική μας σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθούμε 50,5 εκατομμύρια παιδιά και πάνω από 10,5 εκατομμύρια έγκυε και σε γυναίκες και στην Αφρική και στην Ασία. Σε 9 χώρες εφαρμόζουμε ε, τέτοια προγράμματα επισητιστικά που βασίζονται στην ισότητα των ευκαιριών για να δώσουμε σε αυτά τα παιδιά ένα καλύτερο ξεκίνημα για τη ζωή. Επίσης, ανοσοποίηση συμβαδίζει με αυτή την στρατηγική. και Τα νέα εμβόλια συνεπάγονται και μικρότερο κόστος για να φτάσουμε αυτές ε, τις ε, κοινότητες και οι παγκόσμιε ε, εκστρατείε εμβολιασμού για να απαλείψουμε επιτέλου την ε, ε, πολιομιελίτιδα δεν έχουν επιτύχει, δεν μπορούν να επιτύχουν αν δεν ασχοληθούμε με αυτές τις μακρινές κοινότητε και περίπου το 80% των παιδιών τώρα επωφελούνται από αυτά τα εμβόλια αλλά παρόλα αυτά κάθε χρόνο 2 εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν επειδή δεν έχουν αυτό το απλό εμβόλιο. Αυτό φυσικά δεν μπορεί να συνεχιστεί και τώρα ε, ε, ε, ε καλύπτουμε 4 στα 5 παιδιά. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να καλύψουμε 5 στα 5 παιδιά. Ε, η εκπαίδευση είναι ένα άλλο τομής όπου μπορεί να σημειωθεί η πρόοδος και θα έχουμε μεγάλα μερίσματα αν υλοποιήσουμε μια σωστή πολιτική. Ε, ε, γνωρίζουμε ότι η εκπαίδευση είναι ο καλύτερο δρόμο για να απελευθερωθεί από τη φτώχεια μια χώρα και αυτό ισχύει όλο ιδιαίτερα για τα κορίτσια γιατί έτσι θα μπορέσουν να έχουν έναν αξιοπρεπή μισθό, να παντρευτούν, να κάνουν παιδιά και να εξασφαλίσουν την παιδεία των δικών του παιδιών. από το 1900 390 Έχουμε μειώσει ε, τον αριθμό των παιδιών ε, που δεν πηγαίνουν στο ε, σχολείο από τα 113 εκατομμύρια στα 67 εκατομμύρια και η πλειοψηφία ήταν κορίτσια λόγω τη διακριτική μεταχείριση και της ανισότητας ανάμεσα στα δύο φύλλα. Πρέπει να πάμε να βοηθήσουμε τα κορίτσια αυτά να πάνε στο σχολείο, κάθε παιδί πρέπει να είναι στο σχολείο και να αναβαθμίσουμε και την ποιότητα τη εκπαίδευση. Κανένα έθνο δεν μπορεί να ισχυροποιηθεί, να παραμείνει ισχυρό αν δεν γίνει μια τέτοια επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Είναι απαραίτητο να δημιουργήσουμε δικαιότερες ε, ε, ε, κοινωνίες που δεν αποκλείουν κανέναν και όπως είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ δεν είναι η φόρος η ανάπτυξη εκτός και αν είναι δίκαιη και υπηρετεί όλους τους ανθρώπους. Επιδιώκουμε λοιπόν μια αυξημένη ισότητα και κινητοποιούμεθα και σε άλλους τομείς όπως παραδείγματος χάρη την, ε, τις υγειονομικές υποδομές, την καταπολέμηση του AIDS ε, και φυσικά την προστασία των παιδιών ε, σε, στις ένοπλες σειράξεις. Ε, η χρήση και η κατάχρηση των παιδιών από ένοπλες ομάδες είναι κάτι το τερατώδες και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Έχουμε λάβει εντολή από το Συμβόλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να παρακολουθούμε και υποβάλουμε σε ε, για την κατάσταση και επικουρούμε τις κυβερνήσεις, τι προσπάθειε που κάνουν να αποκινητοποιήσουν και να επανεντάξουν στην κοινωνία τα παιδιά που πλήττονται, προσφέροντας ε, συμβουλές, ε, κατάρτιση, εκπαίδευση για να μπορέσουμε να νοικοδομήσουμε αυτές τις κοινωνίες και ε, τα φτωχά παιδιά είναι ακόμη πιο ευάλωτα όταν είναι τόσο κατεπίγουσα η κατάσταση ε, και ε, το, το πεδίο όπου κατεπηγόντως πρέπει να δράσουμε περισσότερο από όλα τα είναι το κέρας της Αφρικής είναι καταστροφική η κατάσταση για τα παιδιά στη Σομαλία, Αιθιοπία και Κένια και όχι μόνο δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων έχουν ήδη πεθάνει και πάνω από 300.000 παιδιά υποφέρουν από οξύ υποσυντισμό ε, επίκειται ε, ο θάνατός τους τις επόμενες εβδομάδες. Ε, το επίκεντρο όμως είναι η Σομαλία όπου 4 εκατομμύρια παιδιά δεν έχουν τα άκρος απαραίτητα στον Νότο, 1,5 εκατομμύρια παιδιά χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια και εκτιμούμε ότι περίπου 200.000 παιδιά στην Σομαλία υποφέρουν από οξύ υποσυτισμό χωρίς αν δεν λάβουν βοήθεια κάτι επιγόντως αυτά τα παιδιά θα πεθάνουν σύντομα. Ε, στις χειρότερα πληττόμενες περιοχές ε, στο κέντρο και στο νότο της ε, Σομαλίας έχουμε αυξήσει τη θεραπευτική αγωγή για τον οξύ υποσυτισμό και παρέχουμε πρόσβαση σε καθαρό νερό. Έχουμε διευρυμένη ε, κάλυψη ανοσοποίησης κυρίως κατά της ε, και επίσης προσφέρουμε διάφορες υγειονομικές υπηρεσίες και διδατικοποιούμε επιχειρήσεις μας. Ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας ε, σήμερα. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δώσει 68 εκατομμύρια, 68 εκατομμύρια ε, δολάρια και ε, έχουν δεσμεύσει και άλλα κονδύλια. Η e CHO έχει ήδη δώσει 30 εκατομμύρια δολάρια ε, και χάρη σε αυτά τα κονδύλια έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις κατεπίγουσες ανάγκες. Ε, προσοχή όμω η κατάσταση στο κέρα τη Αφρική θα επιδεινωθεί. Η κρίση δεν έχει φτάσει ακόμη ε, στο, στο υψηλότερο σημείο της και εάν δεν βελτιωθεί η κατάσταση με τις συγκομιδές, μα περιμένουν χαλεπότεροι καιροί. Δεν θα πρέπει όμω να αποθαρρυνόμαστε. Είναι μια ευκαιρία και μια υποχρέωση για μα να σώσουμε όσο το δυνατόν δυνατόν περισσότερε ζωέ γίνεται. Καθώ κινητοποιούμε του πόρου μα ε, για να αντιμετωπίσουμε αυτή την καταστροφή, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ε, τι επιπτώσει ε, των σειράξεων αλλά και των κλιματικών αλλαγών που θα πλήξουμε περαιτέρω τις πλέον ευάλωτες κοινότητες παρά τις προσπάθειες που θα κάνουμε για να προβλέψουμε, να προλάβουμε και να προετοιμαστούμε για αυτές και δεδομένων των οικονομικών περιορισμών δυσχεραίνεται η κατάσταση έτσι περαιτέρω. Ε, μειώνουμε λοιπόν και εμείς τις δαπάνες μας, αλλά παρόλα αυτά δεν πρέπει να έχουμε χαμηλότερους στόχους σε σχέση με τη διάσωση της ζωής αυτών των παιδιών. Ε, καταφέραμε να περικόψουμε τις δαπάνες χωρίς να καταργήσουμε κανένα πρόγραμμα και ε, πρέπει να ε, καταλάβουμε όλοι ότι κάθε ευρώ μπορεί να βοηθήσει για ένα εμβόλιο, για μια κουνουπιέρα ή για ένα παιδικό βιβλίο Επίσης χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια για να είμαστε υπόλογοι. Το Διοικητικό Συμβούλιο της UNICEF ε, σχάτωσε να μία απόφαση για να επιτρέψει σε διακυβερνητικές οργανώσεις όπως η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και το Παγκόσμιο Ταμείο να έχουν πρόσβαση στις εσωτερικές εκθέσεις ελέγχου της UNICEF και ένα ε, πολύ σημαντικό επόμενο βήμα ε, που επήγεται είναι οι εκθέσεις μας να είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας μέχρι το, έτος, ε, μέχρι το τέλος μάλλον το 2012 ή και νωρίτερα. Αυτό θα είναι κάτω ρηξικέλευθο. Σε όλες τις προσπάθειες που μόλις σας περιέγραψα ε, δηλώνουμε με υπερηφάνεια ότι επιδιώκουμε ε, κοινού στόχου με την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και χωρί ε, συνεργασία και χωρί να εργαζόμαστε με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο δεν θα επιτύχουμε σε αυτέ τι προσπάθειέ μα. Ε, ελπίζω και εσεί να είσαστε περήφανοι για τι θετικέ επιπτώσει τη συνεισφορά σα, όχι μόνο προ τη UNICEF αλλά και προ άλλε οργανώσει, διότι αυτού που υπηρετούμε όλοι είναι τα παιδιά. Ε, προσβλέπουμε στη μελλοντική μα συνεργασία συνεργασία, επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων και πρόοδος ε, προ αυτό που θα έπρεπε να ισχύει, όπω σα έλεγα, ε, προ ένα κόσμο που θα ε, επέλθει. Ένα κόσμο όπου θα ευημερούν τα παιδιά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Λέικ. Πραγματικά πληρέστατη η παρουσίασή σας, συγκινητική και πάρα πάρα πολύ επίκαιρη. Στην συνεδρίαση αυτή συμπροεδρεύει και η συνάδελφος Κρέτσου, η οποία είναι αντιπρόεδρος ε, της Επιτροπής Ανάπτυξης και στην οποία ε, δίνω την Προεδρία και το συντονισμό της συζήτησης. Παρακαλώ κυρία Κρέτσου, ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως ε, και για μένα είναι μεγάλη τιμή να συμπροεδρεύω σε αυτή τη συζήτηση μαζί σας. Εκτιμούμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι είστε εδώ παρόν δεδομένου ότι βιώνουμε και πάρα πολύ δύσκολους και χαλεπούς καιρούς και έχουμε συγκρούσεις ε, σε όλο τον κόσμο. Με τη UNICEF ε, τα τελευταία χρόνια δημιουργήσαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά και με την ευκαιρία των ε, ε, European Development Days το 2010 και μαζί κάναμε πολύ ε, σημαντική δουλειά στη γνωμοδότηση για τα δικαιώματα των παιδιών στην ΑΕΤ. Θα ήθελα να εκφράσω την επιθυμία μας να επεκτείνουμε περαιτέρω αυτή την ήδη καρποφόρα συνεργασία μεταξύ ε, των διοργάνων, διότι γνωρίζουμε ότι οι συνέπειες των ένοπλων σειράξεων πλήττουν κυρίως ε, τα παιδιά και τις γυναίκες. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ε, τι μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε και μια έκθεση για τις γυναίκες και τα παιδιά καιρό πολέμου. Υπάρχουν επίσης και προβλήματα και μεταφοράς ε, παιδιών ε, σε κατάλληλες εγκαταστάσεις και ε, δυστυχώς τα παιδιά αποτελούν και αντικείμενο απάνθρωπων καταχρήσεων. Θα ήθελα να αναφερθούμε και στο θέμα των ομήρων. Ίσως μπορείτε να μιλήσετε λίγο γι' αυτό στο τέλος της παρέμβασής σας. Είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο, ιδιαίτερα στα πρόσφατα γεγονότα της Αραβικής Άνοιξης. Είχαμε πολύ ε, σημαντικά προβλήματα. Υπάρχει επίσης και το ε, θέμα του, της χρήσης των γυναικών που τις υποχρεώνουν να ε, βοηθήσουν ε, πολεμιστές. Επίσης υπάρχει και το θέμα των παιδιών στη Σομαλία τα οποία στρατολογούνται για να πολεμήσουν στην πρώτη γραμμή και εκπαιδεύονται για να κάνουν επεθέσει ενώ ταυτόχρονα του αρνείται το δικαίωμα στην παιδεία. Ε, ξέρουμε ότι ήδη διαστηριοποιείται η UNICEF στη Σομαλία αλλά θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο δραστήριοι, πολύ περισσότερο δραστήριοι στην περιοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία από τους πιο σημαντικούς δωρητές, αλλά δεν διαδραματίζει πάντα τον πιο σημαντικό ρόλο, δυστυχώς, σε ε, περιοχές όπου έχουμε σειράξεις και θα πρέπει να δούμε λίγο και τα θέματα του ποιο είναι υπόλογο σε ποιον. Ε, το θέμα τη διαφάνεια, όπω είπατε κι εσεί, ε, γίνεται όλο ένα και πιο σημαντικό. Οι χώρε γίνονται όλο και πιο εγωίστριε και θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι τα κονδύλια τα οποία δίδουμε φτάνουν στους σωστούς ανθρώπους και πηγαίνουν στο σωστό χώρο εκεί όπου είναι απαραίτητα. Επίσης, από πλευράς Επιτροπής Ανάπτυξης ε, θέλαμε να αναφερθούμε και στα παιδιά στη Μαλαισία. Το 2011 30 παιδιά κρατήθηκαν όμοιροι στη Μαλαισία και θα ήθελα να ξέρω πώς έχει η κατάσταση ε, διότι εδώ και δεκαετίες συνεχίζονται αυτά τα φαινόμενα και επίσης έχουμε και ε, τα γεγονότα στην Ιρλανδία ε, παιδιά τα οποία είναι αντικείμενο κακοποίησης ακόμα και μέσα στα σπίτια τους. Ίσως θα πρέπει να βρούμε λοιπόν νέου τρόπους, συνεργασία και να προσπαθήσουμε να, να αποτρέψουμε συγγνώμη, την επιδείνωση του φαινομένου. Αυτά είχα να πω ως ε, ε, Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ανάπτυξης και τώρα θα ήθελα να ξεκινήσει η συζήτηση και να δώσουμε το λόγο στους ε, συναδέλφους. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από τους συναδέλφους από τις Επιτροπές Εξωτερικών Υποθέσεων και Ανάπτυξης να λάβουν το λόγο. κύριος Παντσέρη, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα και εγώ με τη σειρά μου για την παρουσία του εκτελεστικού διευθυντή της UNICEF διότι πρόκειται για μια σημαντική ευκαιρία διαλόγου και επειδή θεωρώ ότι τα όσα κάνετε είναι αδιαμφισβήτητα ιδιαίτερα σημαντικά είστε άλλωστε άτομο εγνωσμένου κύρους και σεβαστό ανά τον κόσμο και μπορείτε να κινητοποιήσετε ενέργεια και πόρους για να αντιμετωπίσετε τα διάφορα προγράμματα τα οποία μας έχετε αναφέρει. Θα ήθελα παρόλα αυτά να ζητήσω την άποψή σας ε, για το γεγονός ότι δυστυχώς ε, τα θέματα τα οποία μας απασχολούν δεν είναι απλώς και μόνο ανθρωπιστικής φύσεως. Πολλά από τα προβλήματα που καλείστε να αντιμετωπίσετε είναι άμεση απόρρια πολιτικών επιλογών και του γεγονότος ότι επιτρέψτε μου και τον όρο Έχουμε μια θετική κοινωνία η οποία είναι ευρύτατα αφοσιωμένη στην ε, εντατική εκμετάλλευση των πόρων, φτάνοντας μέχρι και την κατάχρηση των πόρων αυτών και καταγγέλλεται συνεχώς ε, ότι σε παγκόσμια κλίμακα τα δύο τρίτα των πόρων κρατούνται από το 1 τρίτο του πληθυσμού και εδώ διαπιστώνουμε στην πράξη ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να κάνουμε μια αξιολόγηση κυρίω πολιτική πέραν της ανθρωπιστικής πτυχής και για τα όσα υλοποιούνται και ως, για τα όσα είχαμε ε, από πλευράς ανάπτυξης τα οποία αποτελούν και πηγή της έλλειψης ισορροπίας. Και μήπως θα έπρεπε η UNICEF να ε, εμπλακεί περισσότερο στο πολιτικό επίπεδο, περισσότερο από όσο συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Τόσο όσον αφορά την αρχική κατάρτιση οποιασδήποτε μορφής παρέμβασης, ε, όσο και όσον αφορά την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Διότι πολλές φορές δίνεται η εντύπωση, μπορεί να ασφάλω εγώ στην αξιολόγησή μου βέβαια, ότι η παρέμβαση γίνεται κατόπιν ορτής και όχι ε, εκ των προτέρων. Τότε δηλαδή που είναι απαραίτητο. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω κατά πόσον θεωρείτε ότι είναι απαραίτητο να συμμετέχετε περισσότερο στις ε, διεθνείς πολιτικές πλατφόρμες ε, και αν θεωρείτε ότι ήδη συμβαίνει αυτό, πώς έχει η κατάσταση, Ιδίω όσον αφορά την μεγαλύτερη δυνατότητα ε, ένταξης των εργασιών σας, ώστε να είναι χρήσιμες ε, όσα κάνετε, όχι μόνο εκ των προτέρων, αλλά και εν είδη πρόληψης. Ευχαριστώ. Κάποιο άλλο, Κάποιος άλλος θέλει το λόγο. Ο κύριος Μπροκ. Mm-hmm. Uh, uh, Οπότε, ε, αφού επιμένετε... Μπορώ, μπορώ να ρωτήσω κάτι αν θέλετε, λέει ο κύριος Μπρόκ. Uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπουμε. Νομίζω πριν από 15 χρόνια είχαμε συναντηθεί πρώτη φορά. Έχω μία ερώτηση. Αυτή τη στιγμή συζητάμε πολύ και πρέπει να κυρώσουμε κάποιες συμφωνίες με χώρες κεντρικής Ασίας όπου έχουμε προβλήματα παιδικής εργασίας και θα ήθελα να ακούσω την άποψη σας τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Ειδικά καθώς πιστεύω πως είναι νομίζω θέμα κοινού ενδιαφέροντος UNICEF και Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και ποιες θα μπορούσαν να είναι οι καλύτερες μέθοδοι συνεργασίας και να έχουμε και κάποια συμβουλή για το πώς μπορεί να εφαρμοστεί κάτι γιατί συχνά στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε κάποιες προδιαγραφές στις συμφωνίες εμπορίου, σύνδεσης κτλ. Αλλά ποτέ δεν παρακολουθούμε, δεν επαληθεύουμε το εάν γίνονται αυτά τα πράγματα στις τρίτες χώρες. Εδώ πέρα λοιπόν θα ήθελα να ακούσω τη συμβουλή σας γιατί δεν παίζουμε επαρκώς τον ρόλο μας. Thank you. I think... Uh, Ευχαριστώ. Νομίζω η κυρία Λοχμπίλερ, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, θα ήθελε να κάνει κάποια ερώτηση. Δεν ξέρω, ο κύριος Λέικ θα θέλει να απαντήσει πριν, στο τέλος. Yes. Yes, maybe the first Mr. Lake to respond to the questions and... Ε, ίσως καλύτερα να απαντήσει πρώτα ο κύριος Λέικ. Yeah. Please. Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και για τις ε, διαφορετικές και ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Ιδιαίτερα με ενδιέφερε η ερώτησή σας η οποία βεβαίως αφορά την ουσία του τι κάνει η UNICEF και τι δεν κάνει. Η UNICEF είναι η μόνη υπηρεσία του ΟΗΕ που μπορεί να εργαστεί αυτή τη στιγμή στην κεντρική και νότια Σομαλία. Είμαστε η υπηρεσία η οποία ε, κάνει εμβολιασμού για την ε, πολιομιελίτιδα σε περιοχή στο Αφγανιστάν που δεν πατάει κανεί άλλο. Η UNICEF ε, σε συνεργασία με την ευρωπαϊκή κοινότητα ε, κατ' ουσίαν δουλεύει για λογαριασμό της κοινότητας σε χώρες ε, που έχουν τεράστιες πολιτικές ε, δυσκολίες και δυσκολεύουν την παρουσία την άμεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως τη Ζιμπάμπου ή άλλες δύσκολες χώρες, πολιτικά δύσκολες. Οπότε είναι τρομερά σημαντικό η UNICEF να διατηρήσει το καθεστώς της ως όχι μόνο μη πολιτική, αλλά να θεωρείται και τέτοια. Από την άλλη, έχετε απολύτως δίκιο, πως είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχωρίσουμε, ειδικά σε ένα μάκρο επίπεδο, το πολιτικό από το μη πολιτικό, γιατί οι πολιτικές αποφάσεις, σωστά σημειώσατε έχουν τεράστιο αντίκτυπο στις ζωές των παιδιών και στο έργο της ε, UNICEF. Οπότε συζητάμε συνεχώς εντός της UNICEF το ποιο είναι το όριο μεταξύ πολιτικού και μη πολιτικού. Και δεν υπάρχει βεβαίω ένα ξεκαθαρό όριο. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να τοποθετούμαστε σε ζητήματα μεταξύ των οποίων και αυτά τα οποία αναφέρατε σε διάφορα φόρα ε, κατά τρόπο να μην φαίνεται πως παίρνουμε το μέρος ε, κάποιου και να μην φαίνεται πως έχουμε στόχο κάποιο πολιτικό αποτέλεσμα παρά μόνο αποτέλεσμα για τα παιδιά. Ε, καταλαβαίνετε τη διάκριση. Και να σας φέρω ένα παράδειγμα. Εγώ ανησυχώ πάρα πολύ και νομίζω όλοι μας ανησυχούμε στη UNICEF για τις αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης και στην Ευρώπη, σε όλο το βιομηχανικό κόσμο και πολύ περισσότερο στις χώρες ε, των G20 και σε πολλές άλλες για την αναπτυξιακή τους πολιτική, που είναι ένα ευρύτερο ζήτημα. Και θεωρώ πως υπάρχει κίνδυνος να ανησυχούν τόσο πολύ για τα βραχυπρόθεσμα ώστε θα επενδύσουν σε μεγάλα έργα υποδομών που είναι ένταση εργασίας για να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και θα παραβλέψουν τη θεμελιώδη σημασία της επένδυσης στον κοινωνικό τομέα, στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στην υγεία, στην εκπαίδευση των λαών τους και ειδικά των παιδιών. Γιατί Εάν σταματήσουν αυτές οι επενδύσεις θα έχουμε σημαντικό αντίκτυπο στον μελλοντική υγεία αυτών των κοινωνιών. Και όπως ανέφερα στις παρατηρήσεις μου δεν μπορούμε, και το δείχνει αυτό η ιστορία, να έχουμε υγιή ανάπτυξη ε, παρά μόνο εάν είναι δίκαιη και ε, αφορά ολόκληρη την κοινωνία μέσω αυτών των επενδύσεων ε, στην υγεία και την εκπαίδευση ολόκληρη την κοινωνία, όχι μόνο τους πιο ε, ε, ευκατάστατους όπου γίνεται η περισσότερη από την κατανάλωση την οποία αναφέρατε. Οπότε είναι ένα ευρύ και πολιτικό ζήτημα όχι μόνο δικαιοσύνης αλλά ζήτημα και λογικής οικονομικής πολιτικής το να επενδύει κανείς στο μέλλον, δηλαδή να επενδύσει στην υγεία και την εκπαίδευση των παιδιών. Και η UNICEF μεταφέρει αυτό το μήνυμα παντού. Και χαίρομαι που μου δίνετε την ευκαιρία να το πω και εδώ. Αυτό σχετίζεται με τις ερωτήσεις επίσης που θέσατε στην αρχή για την ε, τραγική χρήση των παιδιών στις ενόπλες συγκρούσεις, ε, των παιδιών ε, ο ομήρους ε, τη στρατολόγηση που γίνεται στη Σομαλία για την οποία έκανα μια δήλωση πριν από πολλούς μήνες την δολοφονία παιδιών π.χ. δύο παιδιά δολοφονήθηκαν πρόσφατα στην Ιεμένη τις απώλειες που έχουμε στη Συρία και αλλού παιδιών πράγματα αποκρουστικά οι δύο ρόλοι της UNICEF, όπως είπαμε, πρέπει να ε, εξισορροπηθούν αφενός. Έχουμε μία εντολή από το Συμβούλιο Ασφαλείας που αναφέρεται και διευρύνθηκε πρόσφατα στο ψήφισμα 1998 καθώς ε, πλέον ε, θα μπαίνει κανεί σε μια μαύρη λίστα εάν φορολογεί τα, τα σχολεία τους μαθητές. Έχουμε λοιπόν ένα διπλό ρόλο εδώ πέρα. Το πρώτο είναι να παρακολουθούμε και να αναφέρουμε, κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε βεβαίω ε, και όταν μιλάμε για την παιδική εργασία στην Κεντρική Ασία, κάτι το οποίο κάνουμε. Αλλά ένας ρόλος μας είναι να παρακολουθούμε και να αναφέρουμε και μετά να συνεργαστούμε στενά με την είπατε εκπρόσωπο ε, για την παιδική εργασία για να υποβάλει και αυτή τις εκθέσεις της. Αυτή είναι μια λειτουργία. Η άλλη λειτουργία είναι να συνεργαστούμε με κυβερνήσεις για να απελευθερώσουν τα παιδιά που έχουν στρατολογήσει ή να βοηθήσουμε τα παιδιά αυτά όπως το Ανατολικό Κονγκό να επανενταχθεί τα λοιπά και πρέπει να κάνουμε και τα δύο αυτά πράγματα, κατά το οποίο σημαίνει πάντα πως πρέπει να βρίσκουμε μία ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων παρακολούθησης και την δυνατότητα να συνεργαζόμαστε και να φροντίζουμε τα παιδιά εκείνα που έχουν στρατολογηθεί και αναλόγως είμαστε, ε, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι, ο κύριος παγκόσμιο θεματοφύλακας της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και πάντα πρέπει να τα υπερασπιζόμαστε. Και σε πάνω από 150 χώρες και στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική ε, βγάζουμε δηλώσεις ε, και εκθέσεις ε, εξ ονόματος των παιδιών όπου πιστεύουμε ότι παραβιάζονται αυτά τα δικαιώματα. Ταυτόχρονα πρέπει να γίνεται αυτό κατά τρόπο ώστε να μας επιτρέψει να συνεχίσουμε να λειτουργούμε προς όφελος αυτών των παιδιών στις χώρες αυτές. Και αυτό απαιτεί ένα βαθμό ξεκαθαρίς διπλωματίας όπου ξεκαθαρίζουμε πως υπερασπιζόμαστε βεβαίως τις προδιαγραφές και τα δικαιώματα που πρέπει να ισχύουν για τα παιδιά αλλά με έναν τρόπο που θα μας επιτρέψει να λειτουργούμε στις χώρες αυτές ανεξαρτήτως του πολιτικού τους συστήματος ή της πολιτικής της κυβερνήσεως τους για λογαριασμό των παιδιών και αν χάσουμε ποτέ αυτή την ικανότητα θα αποτελέσει αυτό πλήγμα για τα παιδιά γιατί όπως είπα μόνο εμείς μπορούμε να δουλέψουμε σε κάποιες πολύ δύσκολες ε, συνθήκες. Κάτι ακόμα. Νομίζω πως αυτό καλύπτει και τα προβλήματα στη Μαλαισία. Αναφέρατε το ζήτημα της ιδρυματοποίησης των παιδιών που είναι ιδιαίτερα πρόβλημα σε κάποιες χώρες ανατολικότερα από αυτήν στην οποία βρισκόμαστε και πιστεύουμε πως η ιδρυματοποίηση των παιδιών, ειδικά παιδιών σε πολύ νεαρή ηλικία, είναι ευριατή μια παραβίαση των δικαιωμάτων του παιδιού, γιατί αν δει κανεί αυτή την συνθήκη μιλάμε κατ' ουσίαν για το συμφέρον του παιδιού και σε καμία περίπτωση η ιδρυματοποίηση δεν είναι προς το συμφέρον του παιδιού σε σύγκριση με ένα οικογενειακό περιβάλλον ή ένα άλλο περιβάλλον το οποίο θα βοηθήσει να έχουν μια ευτυχή παιδική ηλικία και μια παραγωγική εφηβεία. Νομίζω πως κάλυψα όλα τα σημεία αυτά. Συγκεκριμένα τώρα για την Κεντρική Ασία συνεργαζόμαστε με το Διεθνές Γραφείο Εργασία. Ήμουν πριν από δύο εβδομάδες στην Κυργυζία και αναμένουμε την συνεργασία μας και με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτόπου. Επιτόπου, γιατί είμαστε γενικά σε θέση να δούμε πώς εφαρμόζονται τα προγράμματά μας και βεβαίως ε, είμαστε σε επαφή και με κυβερνήσεις και με επιχειρήσεις για να καταπολεμηθεί, όπως είπα, αυτή η αποκλειστική παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στην κυρία Λόμπ Κίλαρ, πρόεδρο της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για να ολοκληρώσει τη συζήτηση. σα. ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Εγώ έχω αναλάβει να βγάλω τα καταληκτικά συμπεράσματα. Επομένω, καταρχά να σα ευχαριστήσω για την παρουσία σα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για τα όσα μοιραστήκατε μαζί μα. Ε, νομίζω ότι ήταν ε, πολύ ενημερωτική και πολύ εντυπωσιακή η παρουσίασή σας. Ε, εντυπωσιακό διότι ούτως ή άλλως θεωρώ ότι η UNICEF ε, κάνει πάρα πολλά και εσείς ξεκινήσατε ε, λέγοντας ότι θα επικεντρωθείτε στις κοινότητες χαμηλών εισοδημάτων και τις ανάγκες ε, των ε, συγκεκριμένων παιδιών και δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να βάλει ερωτηματικό στο θέμα αυτό. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη δυνατή επένδυση που μπορεί να κάνουμε, διότι το σημαντικό μέρος του πληθυσμού μας είναι τα παιδιά μας και είναι και το μέλλον μας. Και είναι πολύ εντυπωσιακό και αυτό που είπατε υπό άλλη έννοια. Με εντυπωσίασε και ε, με γέμισε και όνειδος κατά κάποιο τρόπο ότι εμείς σας ως ευημερούσα κοιμονία κάνουμε τόσο λίγα και με ελάχιστες επενδύσεις θα μπορούσαμε να κάνουμε πάρα πολλά για να εκριζώσουμε κάποιες ασθένειες επί παραδείγματι ή για να βελτιώσουμε τις συνθήκες διατροφής τους. Και αυτό είναι εντυπωσιακό. Και επίσης ε, ε, εσείς επικεντρωνόσαστε στα, ε, παιδιά, στα δικαιώματα των παιδιών. Εμείς νομίζω στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε ακόμα στο στάδιο του βρέφους, διότι μόλις την Άνοιξη φέτος η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Παιδιών. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε να το αναθρέψουμε αυτό το βρέφος και αναθρέφοντας το βρέφος κατά την ανατροφή του να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε και την εμπειρογνωμοσύνη σας. Ε, στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πάντα σε όλα μας τα ψηφίσματα αναφερόμαστε στο δικαίωμα στην παιδεία. Ε, και θα πρέπει να το επισημάνουμε ότι το να επικεντρωθούμε στα παιδιά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν και κατευθυντήριες γραμμές ε, για τις διάφορες μορφές παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υπάρχει και μια κατευθυντήρια γραμμή για τα παιδιά στρατιώτες και οι... Όσοι εργάζονται επί τόπου από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωσης ε, ελπίζω να μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα για να το βελτιώσουν. Είπατε ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεισφέρουν στη UNOSIF με 68 εκατομμύρια δολάρια στο κέρας της Αφρικής είπατε έτσι, ενώ ε, η Ασία με 30 ε, όλοι κατανοούμε ότι είναι πολύ σημαντικό, είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη να σας βοηθήσουμε και να συνεχίσουμε και τη χρηματοοικονομική υποστήριξη ώστε να μπορέσετε να κάνετε ακόμα περισσότερα. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι για την ε, σημερινή σας παρουσία. Let's start the last uh, point on our agenda. με το τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Μία συζήτηση για μία συνεπή πολιτική έναντι αυταρχικών καθεστώτων. Μία καλύτερη χρήση των περιοριστικών μέτρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το θέμα το 2013 και 14 στην ημερήσια διάταξη. Και προτείνουμε να δώσουμε πρώτα απ' όλα τον λόγο στον κύριο Γκραμ Βάτσον και μετά στην κυρία Πορτέλα. Και μετά θα γίνει μια συζήτηση. Νομίζω πως έτσι θα γλιτώσουμε λίγο χρόνο και θα καλύψουμε τα ζητήματα αυτά έτσι, ολοκληρωμένα. Χωρίς περαιτέρω λοιπόν καθυστέρηση έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην έκθεση αυτή σκοπεύω να χρησιμοποιήσω μία από τις νέες αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου υπό τη μορφή μια σύσταση προς το Συμβούλιο, αν και αντιλαμβάνομαι βεβαίω πώς θα έπρεπε να απευθυνόμαστε προς το Συμβούλιο, την Κομισιόν και την ύπατη εκπρόσωπο, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους. Άλλωστε, η έκθεση αυτή αφορά τις κυρώσεις. Θα γνωρίζετε, κύριε Πρόεδρε, πως δεν υπάρχει ένας κοινό ορισμός των κυρώσεων, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, είναι μάλιστα ε, ένα από τα πιο επίμαχα μέσα εξωτερικής πολιτικής που έχουμε, αλλά ένας βασικός ρόλος και όφελός τους είναι η ικανότητά τους να στιγματίζουν και να απομονώνουν τους στόχους τους. Πάντα εμείς αναφερόμαστε στις κυρώσεις ως περιοριστικά μέτρα και προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε στοχευμένες και έξυπνες κυρώσεις που στοχεύουν άτομα ή ελίτ ε, χρησιμοποιώντας μαύρες λίστες ατόμων γιατί θεωρούμε πως αυτό είναι πιο αποτελεσματικό από συνολικά οικονομικά εμπάργο και πηγαίνουμε πέρα από τις κυρώσεις ε, που συμφωνούνται στο επίπεδο του ΟΗΕ αρκετά συχνά. Όμως δεν έχουμε συνολική πολιτική κυρώσεων ως Ευρωπαϊκή Ένωση παρά το ότι η ε, Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας έχει ζητήσει από την Κομισιόν να δει αυτό το θέμα. Η έκθεση αυτή λοιπόν εξετάζει τις μονομερείς ε, κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι αυτές που απορρέουν από αποφάσει του ΟΗΕ και ζητάει ακριβώς μια συνολική πολιτική για τις κυρώσεις αναγνωρίζοντας πως αυτό έχει επιπτώσεις στους πόρους και πως θα απαιτηθεί από τα κράτη-μέλη να μοιράζονται πληροφορίες με τις αρχές της Ένωσης, παραδείγματο χάρη για το τι βρίσκεται σε τραπεζικούς λογαριασμούς έτσι ώστε να μπορεί να παγώσει. Ένα από τα επιχειρήματα κατά αυτής της έκθεσης θα μπορούσε να είναι πως η πολιτική των κυρώσεων είναι υπομορφή αντίδρασης και όχι πρόληψης. Και έτσι θα μπορούσε να μην επιφέρει αλλαγή καθεστώτος. Η άποψή μου είναι πως ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πάρα πολύ αποτελεσματική στην προώθηση αλλαγής καθεστώτος και μια τέτοια συνολική και προληπτική πολιτική κυρώσεων θα ενισχύσει αυτή τη δυνατότητα της Ένωσης. Μια αντίρρηση στις ε, κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι στιγμής, ε, ένα στόχος, με συγχωρείτε, μέχρι τώρα ήταν το να αποτρέπει κυβερνήσεις αυταρχικών ε, καθιστώτων από τέτοια συμπεριφορά. Σκεφτούμε παραδείγματος χάρη τη Βυρμανία ή την Ζιμπάμπουε ή ακόμα και την ακτή του Ελεφαντοστού. Θα μπορούσε να ρωτήσει κανείς γιατί δεν ε, επιβάλλουμε κυρώσεις σε όλα τα αυταρχικά καθεστώτα όπως παραδείγματος χάρη τη Σιγκαπούρη ή τη Σαουδική Αραβία. Γιατί βεβαίω το να μην εφαρμόζουμε αυτά τα περιοριστικά μέτρα με τρόπο όμοιο βλάπτει την αξιοπιστία της Ένωσης και μειώνει την αποτελεσματικότητα των ίδιων των μέτρων. Δεν ισχυρίζομαι, κύριε Πρόεδρε, πως είμαι ειδικό στο θέμα αυτό. Ευχαρίστω να δεχτώ την Συμβουλή Συναδέλφων και καλωσορίζω τις ε, τροπολογίες τους. Αλλά θεωρώ πως η Ένωση καλά θα έκανε να έχει μια τέτοια συνολική πολιτική. Το εξηγώ και αντιλαμβάνομαι βέβαια πως ε, η επεξηγηματική μου δήλωση θα χρειαστεί κάποια επέκταση θα καταθέσω και εγώ ίδιος δύο τροπολογίες. Η μία αφορά την ενεργοποίηση ρητρών ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διμερείς εμπορικές συμφωνίες και μία η οποία αφορά την δίωξη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσων ξεφεύγουν από αυτές τις κυρώσεις ή προσπαθούν να βοηθήσουν άλλους να ξεφύγουν από τις κυρώσεις. Αλλά η έκθεση αυτή ζητά σαφέστερους ορισμούς του πότε θα πρέπει να εφαρμοστούν τέτοια περιοριστικά μέτρα, ποια θα μπορούσαν να είναι αυτά τα μέτρα, ποιο θα είναι το πολιτικό πλαίσιο στο οποίο τοποθετούνται. Ζητάει επίσης ε, την διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής πολιτικής κυρώσεων, ζητώντας από τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν με τρόπο ενιαίο και αυστηρό αυτές τις κυρώσεις επίσης για να διασφαλίσουμε πως θα έχουμε κάποια συνοδευτικά μέτρα των κυρώσεων για να υπάρχει αυτή η αρχή της εφαρμογής τους και να έχουμε μια συνολικότερη προσέγγιση ε, κομισιών και Ευρωπαϊκής Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Επίσης ζητάει να διαμορφώσουμε μια συνεκτική πολιτική εντός της Ένωσης και να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε διεθνή στήριξη για τις πολιτικές αυτές, ειδικά με στόχους εντός της χώρας την οποία στοχεύουμε. Οπότε θα μπορούσαμε να έχουμε την βάση ε, αυτού του οποίου με κάποιο κίνδυνο θα μπορούσαμε να περιγράψουμε ως εθική εξωτερική πολιτική. Εγώ θα έλεγα μια εξωτερική πολιτική από την οποία δεν απουσιάζει η ηθική και ε, στην οποία εφαρμόζονται τουλάχιστον με τρόπο ομοιόμορφο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πράγματι, δικαίως λέτε πως ε, χρησιμοποιείται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους αυτό το μέσο και ξέρετε πως είναι ούτως ή άλλως μια πολιτική απόφαση η επιβολή κυρώσεων και αυτό δεν σχετίζεται απολύτως με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά το είπαμε χτες στην ψηφοφορία ε, για, τον, ε, για τη Συρία στον ΟΗΕ νομίζω είναι ενδεικτικό το τι συνέβη. Θα ήθελα τώρα λοιπόν να δώσω λόγο στην κυρία Πορτέλα Ευχαριστώ πολύ. Το παρόν ψήφισμα ασχολείται με την ε, συνέπεια των ε, πολιτικών κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από ακαδημαϊκής πλευράς μας ενδιαφέρει το κατά πόσον μπορούμε να πουλήσουμε, να πλασάρουμε καλύτερα στους Ευρωπαίους πολίτες τις κυρώσεις όταν φαίνεται ότι έχουν αποτελέσματα. Δηλαδή δεν επαρκεί ε, να ε, επιβάλλουμε κυρώσεις, πρέπει να έχουν και αποτελέσματα. Γι' αυτό προτείνω τέσσερις μεταρρυθμίσεις. Καταρχάς θα πρέπει να τις καθαρίσουμε καλύτερα. Ε, οι κοινέ αποφάσεις συνήθως εξηλούν τα αίτια ε, και όχι τους στόχους ε, των κυρώσεων και το τι θέλουν να επιτύχουν. Πιο συγκεκριμένα, όταν καθορίζουμε τους στόχους θα πρέπει να δείξουμε και με ποιο τρόπο μπορούμε να μετρήσουμε το αποτέλεσμα των στόχων αργότερα. Δεύτερον, σωστά ζητάμε να μετρήσουμε τα αποτελέσματα των κυρώσεων. Ωστόσο, τα αποτελέσματα των κυρώσεων δεν θα πρέπει να μετρώνται αυτή τη στιγμή έχουν εφαρμοστεί οι κυρώσει, θα πρέπει να εξεταστούν και εκ των προτέρων. Θα πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση αντικτύπου για να ε, σχεδιάσουμε τις κυρώσει κατά τρόπο ώστε να είναι πιο αποτελεσματικέ. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιστοποιήσουμε και το σχεδιασμό των μέτρων και των κυρώσεων που επιβάλλουμε. Αυτό βεβαίω θα πρέπει να περιλαμβάνει και μια εις ανάλυση των κοινωνικών και οικονομικών ε, καταστάσεων των δομών, πώς θα επηρεάσουν κάποιους τομείς της οικονομίας, κάποιες ε, τομείς της κοινωνίας και πώς ε, θα είναι αποτελεσματικά ε, τα μέτρα της ελίτ στη χώρα στόχο. πώς επηρεάζουν την ελίτ ε, ε, και τον πληθυσμό και τι υποστήριξη έχει η ελίτ ε, στην κοινωνία. Επίσης, θα πρέπει να συνοδεύονται και από μια διαδικασία επικοινωνίας με τους επικεφαλείς και τους ηγέτες για να είναι εν γνώση τους το γεγονός ότι πάντα πρέπει να ξέρουν τι να κάνουν ώστε να έρθουν οι κυρώσεις και να γνωρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα άρει τις κυρώσεις αν συμμορφωθούν. Ε, θέλουμε να έχουμε ένα μηχανισμό τακτικής διαβούλευσης ε, και παρακολούθησης και αυτό κάνουμε και στις χώρες ΑΚΕ. Αναφέρομαι στην αναστολή ε, της αναπτυξιακής βοήθειας που έχουμε στο άρθρο 96 των Συμφωνιών Κοτονού και ίσως από τη συμφωνία αυτή θα μπορούσαμε να μεταφέρουμε και το, ε, τις αντίστοιχες στο πλαίσιο των θεμάτων των υπολείπων χωρών. Υπάρχουν δύο τμήματα, ένα στην υπηρεσία εξωτερική δράση και ένα σε ένα άλλο τμήμα. Θα μπορούσαν αυτά να συγχωνευτούν ώστε να υπάρχει καλύτερη συνέργεια και να χρησιμοποιήσει την εμπειρογνωμοσύνη του το τμήμα αυτού. Θα μπορούσε ίσως να χρησιμοποιήσει και εξωτερικούς ε, συνεργάτες για να κάνουν μια αξιολόγηση αντικτύπου πριν και μετά την επιβολή των κυρώσεων. Ευχαριστώ πολύ. Uh, μπορούσαμε βέβαια και αντί για ένα τμήμα να καταλήξουμε σε τρία τμήματα. Συνήθως έτσι γίνεται. Τέλος πάντων, σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι γνωρίζετε τώρα ότι υπάρχουν αρκετοί σκιώδεις εισηγητές ε, για το θέμα αυτό και αρκετοί συνάδελφοι που θέλουν το λόγο. Σας έχω σημειώσει και θα ήθελα να ζητήσω από την κυρία Γέγκερ καταρχάς να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τους δύο προλαλήσαντες και θα ήθελα να τονίσω πως η πρωτοβουλία αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική και καλά θα κάνουμε εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεχίσουμε αυτή την πρωτοβουλία την οποία λάβαμε και Αναφέρθηκε επίσης πως πρόκειται για πολιτικές αποφάσεις, καλά θα κάνουμε να είμαστε και εμείς αυτές τις πολιτικές αποφάσεις. Έχουμε και το δικαίωμα να ζητάμε αυτά τα πράγματα μετά την Λισαβόνα. Έχω κυρίως κάποιες ερωτήσεις που ελπίζω να ξεκαθαρίσουν και ελπίζω να τις ξεκαθαρίσουμε με τροπολογίες. Εγώ δεν βλέπω ένα ξεκάθαρο ορισμό του τι είναι αυταρχικό καθεστώς. Ο εισηγητής, ο κ. Βότσον, είπε πως ε, υπάρχει μια κάποια συνέπεια εδώ πέρα, τι κάνουμε με την χ χώρα και με την ψ χώρα. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Πρέπει να ξέρουμε πάρα πολύ ακριβώς ε, σε ποιο βαθμό θα μπορούσαν να βλάψουν την κοινωνία των πολιτών οι κυρώσεις γιατί ε, θέλουμε να μειώσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις των κυρώσεων στον πληθυσμό και δεν θέλουμε μόνο να ζητάμε και να αποφασίζουμε ε, κυρώσεις αλλά να έχουμε και ένα σενάριο εξόδου και ένα μεταβατικό επίσης. Και θα ήθελα να ακούσω πράγματι εδώ πέρα ποιον ρόλο μπορεί να παίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μπορεί να βοηθήσει τη διαδικασία εξέτασης, στην επιτήρηση των ε, κυρώσεων αυτών ε, ή να βοηθήσει στην εφαρμογή. Κύριε Βότσον, θα σας στήριζα και εγώ στην απέτηση που είχατε να αποτελέσουν βάση οι ρήτρε ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις διμερεί εμπορικέ συμφωνίες. Π.χ. τώρα διαπραγματευόμαστε με το Μαρόκο και στις διαπραγματεύσεις αυτές νομίζω απέχουμε ακόμα. Οπότε πρέπει επίσης να πούμε πως πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Δεν μπορούμε με τη μία χώρα να λέμε πως ε, εμείς ε, ναι εντάξει θέλουμε κτλ και άρα όλα πηγαίνουν καλά ενώ κάποια άλλη χώρα η οποία δεν είναι τόσο φιλική προς τα εμάς να τις επιβάλλουμε κυρώσεις. Πρέπει να έχουμε κάποιες ε, βασικές αρχές. Επίσης βεβαίω δεν θα πρέπει να διακόπτουμε τις σχέσεις με τα κράτη και να υπάρχει παρόλα αυτά ένας διάλογος έτσι ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε την πιθανή μελλοντική δημοκρατική μετάβαση και να διασφαλίσουμε πως η κοινωνία των πολιτών πάντα θα μας ε, βοηθάει εδώ πέρα και θα πρέπει να σκεφτούμε πως θα μπορέσουμε να εγγυηθούμε να μην μετράμε τα κράτη-μέλη με δύο μέτρα και δύο σταθμά, να υπάρξει ένας ξεκάθαρος ορισμός του τι είναι αυταρχικό καθεστώς να ξέρουμε πότε ξεκινάνε οι κυρώσεις, ποιες είναι οι συνθήκες για κυρώσεις, τι θέλουμε, πώς θα τις χειριστούμε και υπό ποιες συνθήκες θα τις σταματήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για αυτή την πρώτη συζήτηση και αναμένω την συνεργασία μας. Της. Κύριο Ζάλα. Ε, ευχαριστώ. Ο κύριος Βάτσον, είπε ότι δεν είναι ειδικό για αυτά τα ζητήματα. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι είναι μια ε, πολύ καλή έκθεση, πολύ καλά δομημένη, έχει εξετάσει διεξοδικά το θέμα, φαίνεται αυτό και θα ήθελα να κάνω λοιπόν τρία σχόλια. Το... Ε, υπάρχει το γνωστό πρόβλημα διαφωνίας ανάμεσα τα κράτη-μέλη. Κάποιο κράτος θα μπορούσε να καλλιεργήσει ε, ε, εμπορικές σχέσεις, να αναπτύξει ιστορικές σχέσεις ε, με, με κάποια τέτοια πολιταρχικά καθεστώτα με τον κόσμο και αυτό υπονομεύει τη δυνατότητα του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιβάλλει με καθολικό τρόπο τις κυρώσεις κατά αυτών των καθεστώτων. Εντοπίζεται το πρόβλημα αυτό μέσα στην έκθεση και στην παράγραφο 1 προτείνεται μία λύση να έχουμε ε, ποσοτικά και πιο αυστηρά σε κάθε περίπτωση κριτήρια για την ε, απόφαση επιβολής ε, κυρώσεων. Φυσικά το πρόβλημα είναι ο ορισμός του πολιταρχικού καθεστώτος όπως είπε ο συνάδελφος αλλά νομίζω ότι είναι σαφής η πρόταση παρόλα αυτά. Δηλαδή, αν είναι, υπάρχουν αντικειμενικά και συγκεκριμένα κριτήρια για να ενεργοποιηθούν οι κυρώσει, θα είναι δυσκολότερο για τα κράτη-μέλη να παρεμποδίσουν αυτή την πολιτική, γιατί συχνά αυτά κάνουν τα κράτη-μέλη. Έτσι θα έχουμε ευρύτερη ε, δράση και δεν θα είμαστε τόσο επιλεκτικοί όπως κάνουμε αυτή τη στιγμή. Εν γέννη συμφωνώ με τον εισηγητή, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το παζάρι που γίνεται εδώ. Δηλαδή, αν γίνουν πιο ε, αυτόματες οι θα χάσουμε την στρατηγική ευελιξία και δεν σημαίνει ότι το ότι θα είμαστε περισσότερο συνεκτικοί στη δράση μας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Αυτό που μας ενδιαφέρει να επιτύχουμε τους στόχους μας. Εξάλλου αυτή, αυτό είναι το παιχνίδι της πολιτικής ε, και των ε, και του κατεστημένου κάθε κράτους. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια ευελιξία για να μπορούμε να χρησιμοποιούμε ε, τις ε, η κυρίως ένα πολύ καλό εργαλείο την ε, υπόσχεση άρσης των κυρώσεων, λειτουργεί καλά με πολλούς δικτάτορες. Ε, τώρα αυτά που είπατε για τον ορισμό του πολιταρχικού καθεστώτος θα δούμε με προσοχή γιατί αν μπορούσε αυτό να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε κάποιους δικτάτορες εντάξει. Επίσης θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις για το θέμα ε, της ε, εισδοχής ε, των φοιτητών στα πανεπιστήμια που προέρχονται από τέτοιες χώρες. Ξέρετε, με αντιβαίνει στην ηθική αυτό, αυτό το μέτρο το λέω καθότι είμαι και ακαδημαϊκός, ε, αρκεί η βίζα. Ε, αν ε, κάποιος δεν έχει τη θεώρηση, δεν μπορεί ούτε να εισέλθει στη χώρα, ούτε να φοιτήσει. Αυτή η πολιτική ακολουθείται εξάλλου και στη ΣΥΠΑ. Αφετέρου, υπάρχουν και κάποιες θετικές πλευρές. Όταν τα παιδιά ε, του δικτάτορα, είτε πρόκειται για παιδιά φιλών ή για ε, παιδιά της ε, κυβερνητικής παράταξης. Μην ξεχνάτε ότι αυτά τα παιδιά είναι στο, στην πρώτη γραμμή των αλλαγών. Δείτε το, τους γιους του Γκαντάφη. Ας μην ξεχνάμε την γενικότερη εικόνα όταν εξετάζουμε τις λεπτομέρειες. η there is a αυτό είναι ένα πρόβλημα. Σε τέτοια πολιταρχικά καθεστώτα αυτοί οι αξιωματούχοι de facto ασκούν προσωπικό έλεγχο ε, των κρατικών υποθέσεων σε πολλές χώρες κυρίως ε, στις χώρες που έχουν πλούσιους ενεργειακούς πόρους, ε, καθώς και στο τραπεζικό σύστημα. Νομίζω θα συμφωνήσει ο εισηγητής ότι η ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βρει ε, ένα τρόπο για να αποτρέψει αυτή τη δράση μέσω των κυρώσεων. Δεν ξέρω, έχω μπερδευτεί λίγο, αλλά είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ίσως θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε και να βρούμε μια διέξοδο. Είναι ένα εξαιρετικά επίκαιρο πρόβλημα. Um, Ευχαριστώ. κυρία Λέζιν. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομη γιατί τα περισσότερα πράγματα που είχα σκεφτεί έχουν καλυφθεί ήδη από τους προλαλήσαντες και τον ίδιο τον εισηγητή και κάποιες από τις ε, σκέψεις μου ή επιφυλάξεις μου αναγνωρίζονται ήδη από την έκθεση αυτή αλλά Όπως είπα το, και για μένα και για άλλους ε, δεν υπάρχουν ε, ικανοποιητικές λύσεις σε ορισμένα πράγματα όπως τους χάρη στον ορισμό δικτατοριών και αυταρχικών καθεστώτων. Μπορεί λοιπόν να είναι αυτό το μέσο αποτελεσματικό αλλά Βεβαίω θα πρέπει να αναλύσουμε τα μέσα αυτά και την επίδρασή του στο γενικό πληθυσμό. Το μέσο αυτό βεβαίως μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο κατάχρησης και θα μπορούσε κάποια καθεστώτα με τα οποία συνεργαζόμαστε καλά ή εμείς θεωρούμε πως έχουν κεντρική γεωστρατηγική σημασία να ενισχύονται και κάποια άλλα για διαφορετικούς λόγους μόνο να υφίστανται κυρώσεις. Αυτό είναι πράγματι ένα πρόβλημα και με ανισχύει πάρα πολύ. Το είπε και ο εισηγητής τι γίνεται με τη Σαουδική Αραβία, τι γίνεται με το Ουσμπεκιστάν, τον Μπαχρέιν. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να βρούμε κριτήρια ορισμού που θα ισχύουν για όλους για το τι είναι αυταρχικό καθεστώς ή δικτατορία και μετά πραγματικά τα καθεστώτα αυτά να τα αναφέρουμε πλήρως για να μην έχουμε τέτοια προβλήματα. Θα σταματήσω εδώ γιατί όλα τα υπόλοιπα τα είπαν οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Thank you very much. Mr. please. Σας ευχαριστούμε, ο κύριος Κέλλον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, μπορώ, δεν μπορώ παρά να συγχαρώ τον συνάδελφο Βάτσον για αυτήν την ε, πρωτοβουλία. Είναι λογική η συνέχεια της Αραβικής Άνοιξης. Νομίζω ότι θα πρέπει να στείλουμε ένα πολιτικό σήμα από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι να είμαστε συνεκτικοί σημαίνει ότι θα είμαστε και αξιόπιστοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί δεν μπορεί να γίνει παγκόσμιος παίκτη, αν ε, δεν έχει συνεκτική δράση στον καθημερινό πολιτικό της βίο δηλαδή. Επίσης είναι θέμα σεβασμού προς την ίδια την Ένωση. Δηλαδή, μας σεβόμαστε αρκετά ώστε να παίρνουμε στα σοβαρά τις αρχές μας ή όχι. Και ο κύριος Βότσον αναφέρθηκε στην ηθική διάσταση και πιστεύω ότι θα έπρεπε να ε, γίνει ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ε, κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Μια τέτοια προσέγγιση θα λειτουργήσει ως ισχυρό κίνητρο για να προωθήσουμε την εξωτερική μας πολιτική, δηλαδή περνώντας ε, μέσω των αντιπροσώπων μα τη υπηρεσία εξωτερικής δράσης ένα ισχυρό μήνυμα προς τις τρίτες χώρες ότι θα πρέπει ε, με σοβαρότητα να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα. Αυτή είναι και η θεραπεία κατά τον, ε, της πολιτικής θεωρίας του διμερισμού των διμερών σχέσεων κατά τη διαστολή με τις πολυμερείς. Έτσι θα είμαστε αποτελεσματικοί αν έχουμε πιο στοχοθετημένες κυρώσεις παραδείγματο χάρη στην περίπτωση της Λευκορωσίας. Το καταφέραμε αυτό, ε, δηλαδή δεν ε, πλήγησαν οι άμαχοι, δεν περιορίστηκε η ελευθερία κινήσεων. Ε, στοχοθετήσαμε τη δράση μας και πλήξαμε την κυβερνός ελίτ. Όπως είπε και ο συνάδελφος Γέγκερ, πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας, αλλά ο φόβος των αντιπίνων ε, και των ανετικών επιπτώσεων της ε, διπλωματίας μας, στις σχέσεις μας με τις τρίτες χώρες μπορεί να αντισταθμιστεί από ε, την νέα όθηση που θα δώσουμε στην πολιτική, γιατί θα είναι μια κοινή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό θα είναι υποφελές όχι μόνο για τις τρίτες χώρες, αλλά και για εμάς τους ίδιους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Μπιτικόφερ τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σκιώδη συζητήτρια για μας είναι η κυρία Κρόνμπεργκ. Αυτήν ε, αντικαθιστώ. Αλλά αυτό το οποίο θα πω είναι μόνο η δική μου η άποψη και όχι οπωσδήποτε η δική της. Εγώ έχω κάποιες δυσκολίες εδώ πέρα με την έκθεση αυτή καθώς ξεκινούν οι συνάδελφοι να απαιτούν ξεκάθαρους ορισμούς. Δεν είμαι σίγουρος πώς στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής μπορούμε να ξεκινήσουμε να έχουμε ορισμούς και έτσι θα επιτύχουμε κάτι. Ε, αυτό καλό είναι να τα αφήσουμε αλλού. Πρέπει στην εξωτερική πολιτική να είμαστε σε θέση να κρίνουμε τις συγκεκριμένες συνθήκες της συγκεκριμένης περίπτωσης και αναλόγως να ζυγίσουμε τα πράγματα. Και εάν γίνει αυτό και επιτραπεί, τότε δεν έχει κάποια αξία. Και από την άλλη, αν είναι τόσο στενή ώστε αποκλείουν άλλες περιπτώσεις, τότε δεν είναι πρακτική. Οπότε θεωρώ πως το να έχουμε ορισμούς δεν θα καταφέρουμε για να αντιμετωπίζουμε όλες τις περιπτώσεις με τον ίδιο τρόπο δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Εδώ πέρα διαφωνώ κύριε Κέλαμ. Λέτε πως ε, η συνέπεια είναι βασικό κομμάτι του να είναι κανείς παγκόσμιος παίκτη. Η ΕΠΑ το αντίθετο. Η Σοβιετική Ένωση το είχε αποδείξει Κίνα επίσης και εμείς οι ίδιοι στο πλαίσιο του ΟΗΕ πάρα πολλές φορές έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Σωστή η κριτική στα δύο μέτρα και δύο σταθμά, αλλά δεν θεωρώ πως αυτό θα λυθεί με ορισμούς. Αντιθέτως θα πρέπει να συζητάμε κάθε φορά. Δεύτερον, το θέμα των αθαρχικών καθεστώτων και τι σημαίνει αυτό και των ηγετών. Πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ αθαρχικών καθεστώτων και δικτατοριών. Που πολιτική σκοπιά έχει κάποιο νόημα και εγώ δεν θα ήθελα να τα βάλουμε όλα σε ένα καλάθι τι είπα να πει αυταρχικό, περισσότερο αυταρχικό, δικτατορικό κτλ. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Για να τα καλύψουμε με τη μία. Τρίτον, στο VW και X στα σημεία αυτά όπου λέγεται το τι συνέπειες θα πρέπει να έχουν οι κυρώσεις. Κοιτάξτε, μα εδώ πέρα ήδη προτείνουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τους συγγενείς και να λέμε φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τους ηγέτες αυτούς. Δεν μπορούμε να τιμωρήσουμε τους ε, συγγενείς αν ο αδερφός κάποιου ζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μιλάει στον αδερφό του, το δικτάτορα. Δεν ξέρω βεβαίως να συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά θα μπορούσε. Δηλαδή μόνο και μόνο η συγγένεια δεν μπορεί να οδηγήσει στο να λέμε «Α, θα σε τιμωρήσουμε», δεν είναι σωστό. Και τέλος, θεωρώ πως το παρακάνουμε με αυτό το οποίο βλέπω εδώ πέρα στο σημείο αυτό που μιλάει για coercive diplomacy. Θα πρέπει βεβαίω να επιδείξουμε μια συνέπεια όσο γίνεται, αλλά το να λέμε πως η Ευρώπη θα έχει τη δυνατότητα να ασκήσει και βία ή, διπλωμα... ή δηλαδή μια διπλωματία καταναγκαστική όπως τη λέτε εδώ πέρα, ε, μην τα παραλέμε τώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούμε να ασκήσουμε μια κάποια επιρροή, αλλά για coercive διπλώμαση δεν το βλέπω. Ευχαριστώ. Πράγματι, πρέπει να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ κάποιων κεντρικών αρχών που θα μας προσδώσουν την αξιοπιστία στην οποία αναφερόμαστε, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να αφήσουμε και κάποια ευελιξία, διότι υπάρχουν διαφορετικές περιπτώσεις. Ε, και νομίζω ότι ο εισηγητής ε, είναι αυτός ο οποίος θα πρέπει να βρει ποια είναι η διαχωριστική γραμμή μεταξύ των ε, προσεγγίσεων που και οι δύο έχουν αρκετά ωφέλη. Ο κύριος Αλαβράκος παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ο Λόρδος ε, Γκράχαμ Γουάτσον ε, είναι φίλος μου και είναι από τους ανθρώπους εκείνους που ό,τι και να μου έφερνε ένα κείμενο να το υπογράψω χωρίς να το διαβάσω θα το υπέγραφε. Ε, Εποκειμένου έκανα ε, τον κανόνα και το διάβασε. Και με ικανοποιεί ιδιαίτερα η πρόταση του κυρίου Βάτσον για αύξηση της διαφάνειας, για καλύτερο συντονισμό μεταξύ κρατών μελών της Ένωσης, ώστε να εκφράζεται με μία φωνή πάνω σε αυτό το θέμα και έτσι να μην πλήττεται η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών για την κατοχή περιουσιακών στοιχείων ηγετών αυταρχικών καθεστώτων επί του εδάφους. Έγινε συζήτηση για τα αυταρχικά καθεστώτα και εγώ είμαι με την άποψη, συντάσσουμε με την άποψη αποφυγής των ορισμών. Δηλαδή, όταν ορίσουμε τι είναι αυταρχικό καθεστώς, πρώτον θα δώσουμε στα αυταρχικά καθεστώτα την δυνατότητα να παρακάμψουν αυτό τον ορισμό, διότι θα εφεύρουν τρόπους ούτω ώστε να μην εμπίπτουν στις διαδικασίες αυτές και δεύτερον θα περιορίσουμε τη δική μας αντίληψη των πραγμάτων. Παραδείγματο χάρη, δεν μπορώ να αντιληφθώ ότι η έλλειψη ορισμού οδήγησε τη London School of Economics να δέχεται χρηματικά ποσά και χρηματικές ενισχύσεις από τον Καντάφη. Όταν ξέραμε τι είναι ο Καντάφη. Όλη η ανθρωπότητα ξέρει τι είναι ο Καντάφη και πώς ο Καντάφη ταλαιπώρησε την ανθρωπότητα με τον α ή β τρόπο και προκάλεσε την ανθρωπότητα. Βεβαίως με τα κριτήρια τα καθαρά νομικά ο Καντάφη ήταν εκλεγμένο. Εκλεγμένο ήταν βεβαίω και ο Χίτλερ. Εκλεγμένοι είναι πάρα πολλοί δικτάτορε που κατά καιρού έχουν παρουσιαστεί και πάρα πολλοί οι οποίοι κατά καιρού έχουν ασκήσει την εξουσία για κάθε υπέρβαση τη εξουσία του. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι μόνη η εκλογική διαδικασία δίνει την νομιμοποίηση και τον αποχαρακτηρισμό ενός αυταρχικού καθεστώτος. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί βεβαίως και πιστεύω ότι όσον αφορά ε, την ε, επιβολή οικονομικών κυρώσεων κατά τους κανόνες του διεθνούς δικαίου ακόμη και υπό το καθεστώς της συμβάσεως της Λισαβόνος φοβούμαι ότι αυτό είναι πολιτική απόφαση που εντάσσεται στους όρους της αρχής επικουρικότητος. Τι μπορούμε να κάνουμε εκεί. Πιστεύω ότι εκεί θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα συντονισμό των κρατών μελών ει τρόπον ώστε να ασκείται κατά το μάλλον και ήτον μια σαφής πολιτική διαλογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία και έστω χωρίς να είναι ουσιαστική θα παράγει αποτελέσματα λόγω του κύρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της καθιερώσεώς της στα διεθνή πράγματα. Ε, δεν θα ήθελα να κουράσω περισσότερο. Βλέπω τον προβληματισμό του εισηγητού πάνω στο θέμα και βλέπω και τον προβληματισμό όλων μας. Είναι ένα θέμα που ε, έχει φωτιά, είναι κάρβουνο. Είτε το πιάνεις ε, ε, χωρίς να είναι αναμένο σε λερώνει, είτε αν το πιάσεις καμένο σου καίει το χέρι. Αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να δούμε και το άλλο θέμα. Μιλάμε για τεράστια εκατομμύρια τα οποία διακινούν αυτοί οι αυταρχικοί τύποι που παριστάνουν τους ηγέτες των χωρών. Πρέπει να ξέρετε ότι αυτό, αυτό το ποσό το οποίο αφαιρούν από το κράτος τους, το αφαιρούν από το ΑΕΠ της περιοχής στην οποία νηγούνται, εντός ή εκτός εισαγωγικών. Και αυτό το ποσό εντάσσεται σε ένα αργούν κεφάλαιο το οποίο ανατρέπει τις οικονομικές ισορροπίες παγκοσμίω, διότι μιλάμε για τεράστια ποσά. Θυμάστε τι είχε γίνει με τον Μάρκο των Φιλιππίνων, τι ποσά μιλούσαμε και βλέπω εδώ στην αιτιολογική έκθεση για τι πόσα μιλάμε. Πρέπει να δούμε ότι το παγκόσμιο ΑΕΠ με τα στοιχεία του 2009 ήταν 60 τρισεκατομμύρια περίπου δολάρια. Αντίστοιχο είναι το δημόσιο χρέος. 60-59 τρισεκατομμύρια με στοιχεία του 2009 είναι το παγκόσμιο δημόσιο χρέος. Παράλληλα όμως τι υπάρχουν. Υπάρχουν χίλια τρισεκατομμύρια οι καταθέσεις της τράπεζας, η άθληση των καταθέσεων ιδιωτών στις τράπεζες ή εταιριών τα οποία αργούντα κεφάλαια. Από τα 1.003 εκατομμύρια ένα μεγάλο ποσοστό του 30% προέρχεται από, αυτούς, από αυτά τα αυταρχικά καθεστώτα. Δηλαδή μιλάμε για 300 τρισεκατομμύρια δολάρια τα οποία βρίσκονται εκτός νομισματικής κυκλοφορίας και εκτός ε, παραγωγικής διαδικασίας. Πρέπει να μας προβληματίσει πολύ ουσιαστικά το θέμα εάν θέλουμε να διατηρήσουμε τη σοβαρότητά μας η οποία τον τελευταίο καιρό και εν ώψη της άνοιξης της αραβικής έχει τρωθεί διότι από τόμους εκείνοι με τους οποίους συνεργαζόμαστε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση ήρθαν να κατηγορηθούν από εμά σαν αυταρχικοί. Μα μέχρι προχθές τους φέρναμε και τους κάναμε δεξιώσει. Δεν είχαμε καταλάβει μέχρι την πλατεία ε, Ταχρήμ ότι υπήρχε αυταρχικό καθεστώς στην Αίγυπτο. Δεν είχαμε καταλάβει ότι ο Καντάφη ήταν ένας αυταρχικός ηγέτης. Λοιπόν, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δακτυλό μας, πρέπει να φερθούμε πολύ σοβαρά και να μιλάμε πολύ σοβαρά και τι είναι σοβαρό, ό,τι είναι αληθές. Και το αληθές το ξέρουμε όλοι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ τα συχνότερα φαινόμενα είναι να, οι καλοί να γίνονται κακοί. Το λιγότερο συχνό είναι κάποιοι που είναι κακοί να γίνονται καλοί. Και σπανίως κάποιος που είναι κακός γίνεται καλός και μετά ξαναγίνεται κακός και ξανά καλός. Ε, νομίζω ότι εδώ έχουμε φτάσει στο ανώτατο όριο. Δεν μπορούμε να έχουμε κάτι παραπάνω. Κύριος Κασουλίδης παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα ήθελα να σας πω ότι η πρωτοβουλία και η προσπάθεια που έκανε ο κύριος Βότσον είναι αξιέπαινα. Διότι, αντλώντας διδάγματα από την Αραβική Άνοιξη, διερωτάται κανείς πώς όταν η Σοβιετική Άνοιξη κατέρευσε και οι χώρες της Σοβιετικής Ενώσεως απελευθερώθηκαν και στις χώρες της Λατινικής ε, Αμερικής ε, η μία μετά την άλλη οι δικτατορίες κατέρευσαν και αποκαταστάθηκε η δημοκρατία και στην αραβικό κόσμο ε, η χειραφέτηση των γυναικών, τα δικαιώματα των παιδιών δεν είχαν επιτευθεί μέχρι να ε, εξεγερθούν οι λαοί των χωρών αυτών. Ποτέ δεν πολεμήσαμε εμείς για την πραγματική δημοκρατία σε αυτό το τμήμα του κόσμου. Η απάντηση λοιπόν βρίσκεται εδώ. Βρίσκεται στο επεξεγηματικό σημείωμα του κυρίου Γότσον. Τα πετροδολάρια ήταν αυτά τα οποία μας οδήγησαν να έχουμε μάτια ερμητικά κλειστά σε αυτό τον ε, ε, καθόλου αντιδημοκρατικό κόσμο. Ζητώ λοιπόν από τους συναδέλφους να απαντήσουν ειλικρινά στους εαυτούς τους το ερώτημα. Ε, αυτό έχει σημασία να λέμε ποιος είναι αυταρχικός και ποιος δεν είναι. Πριν από ένα χρόνο θα είχαμε συμπεριλάβει τον κύριο Μουμπάρακ ή τον Ζινεντίν Βεναλή σε αυτό τον κατάλογο των αυταρχικών καθεστώτων ε, που θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνουμε σε αυτές τις κυρώσεις. Θα ήθελα πραγματικά να, να αναρωτηθείτε ειλικρινά. Είχαμε καμία πρόθεση να συμπεριλάβουμε αυτούς τους ανθρώπους σε αυτό τον κατάλογο. Λοιπόν, φρονώ ότι θα πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ ε, κυρώσεων που επιβάλλονται μετά από ένα γεγονός, post facto, και περιοριστικά μέτρα, όπως ονομάζονται, για αυταρχικούς ηγέτες, για τις οικογένειές τους και τους απογόνους τους. Και εδώ νομίζω ότι χρειάζεται ένας κώδικας δεοντολογίας, όχι κυρώσεις. Ένας κώδικας δεοντολογίας σημαίνει ότι αν εμεί έχουμε τράπεζες στην Ευρώπη και όταν τους δώσουμε οδηγίε να γνωρίζουν ποιοι είναι οι πελάτες τους για την καταπολέμηση της ε, ε, νομιμοποίησης παρανόμων εσόδων, ε, εάν δεν τηρήσουμε τους κανόνες, ε, ε, έχουμε ξέπλυμα χρήματος. Ουσιαστικά ξεπλένουν τα χρήματα της χώρας τους και τα βάζουν στους προσωπικούς τους λογαριασμούς ή στους λογαριασμούς των οικογενειών τους. Σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει κώδικας διοντολογίας, επίσης και διαφάνεια σε ακαδημαϊκές έδρες ή και σε άλλους οργανισμούς, παραδείγματος χάρη φιλανθρωπικά ιδρύματα, διότι ακόμα και εκεί υπάρχει τρόπος ε, ε, νομιμοποίησης παρανόμων εσόδων που καταλυστεύουν από τους λαούς τους. Ένα κώδικα δεοντολογίας επίσης για τις ποδοσφαιρικές ομάδες. Μια άλλη μορφή, ένας άλλος τομέας ε, στον οποίο ε, χρηματοδοτούν οι δικτάτορες αυτοί. Θα πρέπει να ε, συμφωνήσουμε λοιπόν να υπάρχει ένας ε, κώδικας διοντολογίας για όλους εκ των προτέρων και μετά, όπως είπε και κάποιος συνάδελφος, ε, θα πρέπει να έχουμε εργαλεία τα οποία θα μας επιτρέπουν να απαντούμε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, σε συγκεκριμένα θέματα για συγκεκριμένους δικτάτορες. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν μιλάμε για πετροδολάρια, ξέρετε θυμήθηκα αυτό που είχε πει ένας αυτοκράτορα, αυτοκράτορας πως ε, το χρήμα δεν μυρίζει. Ίσως τα συγκεκριμένα αυτά δολάρια μυρίζουν. Και, και η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά επίση. Οπότε και το ξέπλυμα του χρήματο δεν είναι τόσο κακό. Say, but, uh, Θα έλεγαν κάποιοι. Εν ο κύριο Παντσέρη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα μικρό προήμιο καταρχάς. Στι διεθνέ σχέσει η ευελιξία αυτή καθεαυτή δεν είναι λόγος για να είμαστε συνεπεί. Και εδώ κατά κάποιο τρόπο κάνουμε μία προσπάθεια, μία απόπειρα να ε, βγάλουμε από τη ε, ε, μέση τη Realpolitik. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα στο ίδιο καζάνι, διότι αλλιώς δεν θα έχουμε αποτελεσματική διεθνή πολιτική. Τα όσα έκανε ο συνάδελφος Βότσον νομίζω ότι αποτελούν καλό προήμιο, μπορούν να είναι μια καλή συνεισφορά, ένα σημαντικό σημείο αναφορά για να εφαρμόσουμε μια εξωτερική πολιτική η οποία θα είναι ενιαία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να κάνω κάποιες ε, σύντομες παρατηρήσεις. Επαληθεύοντας και με τον κύριο Βότσον κατά πόσον μπορούμε να βρούμε και σημεία επαφή από ε, αυτόν. Θα ήθελα να μου πείτε καταρχάς αν μπορούμε να βρούμε μία λύση για τον ορισμό του αυταρχικού κράτους. Αν θα μπορούσαμε να έχουμε ένα σημείο αξιολόγησης το οποίο να προβλέπει ένα σταθερό και ένα πιο ελαστικό τμήμα. Δηλαδή, εάν έχουμε ένα ελάχιστο ε, πρότυπο και να καθορίσουμε ένα επίπεδο πέραν του οποίου ξεκινούν οι κυρώσεις και ένα δεύτερο τμήμα το οποίο σχετίζεται με την ελαστικότητα την οποία θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σε περίπτωση που ε, δεν ε, ε, υπάρχει αντίκτυπος σωστός σε σχέση με τις κυρώσεις που επιβάλλονται. Επαναλαμβάνω να υπάρχουν ένα ελάχιστο πρότυπο γιατί δεν μπορούμε να καθορίσουμε το ανώτατο για διάφορους λόγους. Δεύτερον, Θεωρώ ότι υπάρχει ανάγκη να εμβαθύνουμε περισσότερο στο θέμα της αποτελεσματικότητας και της έλλειψης αποτελεσματικότητας των κυρώσεων. Αποτελεσματικότητα αφενός ε, για να ε, μην υπάρχει μια δεσποτική ε, κατάσταση λόγω δεσποτικού καθεστώτος σε μια χώρα και επίσης διότι πολλές φορές διαπιστώσαμε ότι δεν ελήφθη υπόψη ο λαός και ορισμένες φορές επιβάρυναν χωρίς λόγο κάποιους λαούς, ενώ σε κάποιες άλλες ε, περιπτώσεις απλώς γαργάλισαν τα αυταρχικά καθεστώτα χωρίς να έχουν πραγματικό αποτέλεσμα. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε κατά πόσον είναι δυνατόν να κάνουμε μια απόπειρα να συνδυάσουμε αυτό το σημαντικό έργο με τα όσα γίνονται με τις αλλαγές στην πολιτική γειτονία. Διότι το θέμα της ε, ε, αναλογικότητας θα πρέπει να ε, συνδυαστεί και με τις κυρώσεις. Δεν θα πρέπει να είναι δύο εκδιαμέτρου αντίθετες ε, δράσεις, διότι φαίνεται να μην είμαστε συνεπείς και ενώπιον των εταίρων μας. Τέλος, για να απαντήσω σύντομα και στον κύριο Κασουλίδη, εμείς πρέπει, επειδή ακριβώς κάνει καλή δουλειά ο κύριος Βότσον, να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε λίγο το ρόλο και των διπλωματικών μας ε, ε, δυνατοτήτων ανά τον κόσμο να μην περιορίζονται απλώς σε δεξιώσεις και σε επαφές με τα περιτροπής καθεστώτα, αλλά να πηγαίνουν πραγματικά στις χώρες στις οποίες έχουν τοποθετηθεί και θα είχαν αντιληφθεί ίσως κάποιους μήνες νωρίτερα ότι ο Μπεναλή ήταν ε, της κατηγορίας και της υποστάθμης που ήταν. Θα πρέπει να επισκέπτονται ε, λοιπόν λίγο τις χώρες, να μην φτάνουν ως ε, εξωγήινοι στις χώρες και να μην τις μαθαίνουν καθόλου. Θα πρέπει ίσως λοιπόν να το συνδέσουμε και με τις διπλωματικές μας έδρας, να τροποποιήσουμε λίγο το ρόλο τους, διότι θα μπορούσαν να είναι οι πρώτοι που θα αντιληφθούν την κατάσταση σε μια συγκεκριμένη χώρα και να μπορούν αντικειμενικά από εκεί και πέρα να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις τα όσα αποφασίσουμε να εφαρμόζονται εις βάθος. Ευχαριστώ. Uh, Νομίζω ότι ξέρετε ότι αν θέλουμε κάποιο αυτόματο χαρακτήρα, χρειαζόμαστε και ένα κώδικα δεοντολογίας. Εάν δεν τηρηθεί, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα ένα σύστημα επιβολής κυρώσεων. Νομίζω ότι θα λειτουργούσε λογικά ένας μηχανισμός εκτάκτος, κύριε Μπιουτικόφρη, γιατί δεν προβλεπόταν Και μετά θα ακούσουμε τον κύριο Κουκάν και κατόπιν τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά τους δύο εισηγητές για να συνοψίσουν τη συζήτηση. Ευχαριστώ για τη γενεοδορία σας. Να απαντήσω τον κύριο Κασουλίδη λίγο. Ναι, εγώ θα έλεγα πως ε, πράγματι πριν έξι μήνες, ένα χρόνο θα λέγαμε και είχαμε πει πως ο Μπεναλή είναι αυταρχικός και ο Μουμπάρακ. Α, δεν ήταν δύσκολο να να το δούμε. Το θέμα το οποίο... Και εγώ δεν έχω και δυσκολία σήμερα να πω πως ε, και ο Πούτιν είναι αυταρχικός ε, ηγέτης και αυτό το βλέπουμε. Το θέμα είναι το τι κάνουμε μετά από αυτό. Και αν δούμε το σημείο α εδώ πέρα, να αναπτυχθούν σαφή κριτήρια για το πότε θα εφαρμοστούν περιοριστικά μέτρα. Εδώ πέρα πρέπει να πω μια στιγμή για εμένα με το στο θέμα αυτό παίζει ρόλο και η αποτελεσματικότητα ενός μέτρου. Δεν μπορώ έναντι του Χουτζιντάο να κινηθώ με τα ίδια μέσα όπως έναντι του χύψη Αφρικανού δικτάτορα. Δεν είναι ρεαλιστικά το ίδιο πράγμα και αν έχουμε έναν κατάλογο, εάν θέλετε, μέτρων ε, των οποίων περιφέρουμε, ε, δεν είναι αυτή ρεάλ πολιτική, απλά γινόμαστε καταγέλαστοι. Και αυτό δεν το θέλω. Και δεν νομίζω πως το θέλει και ο κύριος Βάτσον. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε κάπως πιο ευέλικτοι στη λύση που θα βρούμε. Ευχαριστώ. Ε, όσο πιο Όσο πιο ακριβή είναι κανείς, τόσο μετά πιο πολύ δεσμεύεται από αυτά τα οποία είπε. Λοιπόν, ο κύριος Κόκαν και μετά ο κύριος ε, Κασουλίδη, πάλι όλος εξαιρετικός. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύντομα και εγώ, Καθώ καθώς ε, όλοι εξέφρασαν όλες τις πιθανές απόψεις. Αυτό το οποίο λέει ο κύριος Γκρέιμ είναι πάρα πολύ καλή καθοδήγηση ε, για την μελλοντική μας. Και βεβαίως μπορούμε να έχουμε κάποιες τέτοιες κατευθυντήριες γραμμές εάν τις σέβονται όλα τα κράτη-μέλη. Εγώ θυμάμαι πως στο παρελθόν η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε υιοθετήσει διάφορες συστάσεις όσον αφορά την Κούβα δεν ε, τις ακολούθησαν όλα τα κράτη-μέλη αυτές τις ε, συστάσεις και όμως αυτά τα καθεστώτα εκμεταλλεύονται πάρα πολύ δεξιοτεχνικά τις ε, διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Όσον αφορά τώρα αυτά τα οποία μας λέει και η έκθεση του Γκάιαμ, πρέπει να εκμεταλλευτούμε πλήρως την εμπειρία της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης στην αξιολόγηση της ε, δυνατότητας επιβολής κυρώσεων και μετά στον συντονισμό αυτών των κυρώσεων. Οπότε θα άξιζε να υπάρχει μια μονάδα εντό υπηρεσία εξωτερική δράση για το θέμα των κυρώσεων. Τώρα για τον ορισμό του αυταρχικού καθεστώτος. Εκεί πέρα είμαι πολύ επιφυλακτικό. Δεν είναι εύκολο να ορίσουμε ένα αυταρχικό καθεστώς. Και εάν συμφωνούσαμε ποτέ σε κάποιον ορισμό, θα ανακαλύπταμε πως ε, θα εμφανίζονταν ένα καθεστώς που δεν τέριαζε ακριβώς σε αυτόν τον ορισμό. Και τι θα κάνουμε τότε. Πρέπει να είμαστε σε θέση να αντιδράσουμε σε οποιαδήποτε κατάσταση η οποία θα προκύψει με τρόπο υπεύθυνο χρησιμοποιώντας τα κριτήρια τα οποία έχουμε στις ε, συστάσεις. Ακόμα και αν είχαμε κάποιον ορισμό θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε ένα υπόδειγμα το οποίο θα μας επέτρεπε να πούμε πως το καθεστώς Α εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία, ενώ το καθεστώς Β όχι. Δεν νομίζω πως θα ήταν χρήσιμο. Σας ευχαριστώ. Κύριε Κασουλίδη, μισό λεπτάκι. Βεβαίω, κύριε Πρόεδρε. Να πω πως αυτά τα οποία είπα για το εάν θα είχαμε συμπεριλάβει το Μουμπάρακ και τα λοιπά, τα είπα σε ένα πνεύμα αυτοκριτικής. Συμπεριέλαβα και τον εαυτό μου. Ε, οπότε δεν ανέμενα κάποια αντίδραση. Και εξάλλου, εγώ συμφωνώ με αυτό το οποίο είπατε κύριε Μπιουτικόφερα όσον αφορά δε την ε, Κομισιόν και την Υπηρεσία εξωτερική Δράσης το Συμβούλιο αποφάσισε κάποιε ρήτρε περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περί αναστολής οποιασδήποτε συμφωνίας ελευθέρου εμπορίου, σύνδεσης οικονομικής συμφωνίας ακόμα και με χώρες με Ε, αδιάκοπη δημοκρατική παράδοση. Μάλιστα. Θα δώσουμε τώρα τον λόγο στον κύριο Ρότζερ Μάθιουζα από την ε, ε, αρμόδια μονάδα της Κομισιόν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση αυτή τη έκθεση. Ναι, Ενέχει κάποιε πολύ χρήσιμε συστάσει και μα βοήθησαν πολύ και τα σχόλια των συναδέλφων που ακούσαμε. Ε, οι κυρώσει ε, υπήρξαν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο ε, στο δεύτερο εργαλειοθήκη τη κοινή πολιτική και πολιτική Άμυνα και έχουν χρησιμοποιηθεί και στα πλαίσια τη Αραβική Άνοιξη και αλλού και φυσικά έχουμε έναν ενεργό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουμε, θα ε, υποβάλουμε ένα σχέδιο κανονισμού και θα μεριμνήσουμε στη συνέχεια για να εφαρμοστεί ομοιόμορφα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημαντικό είναι ο ρόλο τη Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, ε, που επίση ε, προετοιμάζει ένα σχέδιο για ένα μηχανισμό κυρώσεων. Ίσως σας ενδιαφέρει να μάθετε ότι η Πολιτική Επιτροπή του Συμβουλίου ανέθεσε στην ε, ομάδα Ρελέξε του Συμβουλίου να εξετάσει μία σειρά ζητημάτων σχετικά με το χειρισμό των κυρώσεων από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Όλοι θα συμβάλλουμε σε αυτή τη συζήτηση και από αυτή την πλευρά πιο συγκεκριμένα μας βοηθάει το σχέδιο έκθεση ε, του εισηγητή καθώς και οι συστάσεις ε, που κάνει είναι εξαιρετικά επίκαιρες. Ε, θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια αυτού του διαλόγου. Σε αυτό το στάδιο θα ήθελα να σας πω ότι σημειώνουμε όλες αυτές τις παρατηρήσεις και θα λάβουμε σοβαρά υπόψη τις συστάσεις που ανέχει η, έκθεση. Ευχαριστούμε τώρα από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ο, κ. James Key Bright μια σύντομη παρέμβαση. Ευχαριστώ πολύ να συμφωνήσω με τα σχόλια του συναδέλφου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλωσορίζουμε και σημειώνουμε την έκθεση. Μπορεί να σας ενδιαφέρει ε, το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη ζήτησαν ε, μια επιπλέον συνεδρίαση για να προχωρήσει το θέμα ε, συμπεριλαμβανομένης και της εφαρμογής των κυρώσεων ε, θα λάβουμε υπόψη εκεί την έκθεση και χαιρετίζουμε τη σημερινή συζήτηση. Ευχαριστώ. Γκράχαμ για να ολοκληρώσουμε και μετά οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τις κυρίες Γέγλε και Ελένη και τον κύριο Μπιουτικόφερ, την κυρία Γέγλε για το ερώτημα σας και την ε, κυρία Ελένη για τις ανησυχίες σας και το ότι μας συνθυμίσατε την πιθανή κατάχρηση αυτής της πολιτικής. Κύριε Μπιουτικόφερ, πολύ σωστά υπερασπίσατε τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά πολύ ωραίο τρόπο και βεβαίως είχατε και κάποια γνωστά σε όλους μας προβλήματα τώρα. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ρεαλιστή και φονταμεταλιστή Εντάξει, εσείς είστε από ό,τι φαίνεται ρεαλιστής όπως άλλωστε και η κυρία Κρόνμπερκ. Κύριε Παντσέρη. Ευχαριστώ και για τη δική σας παρέμβαση και κυρίως για αυτό που είπατε τη σημασία του να σκεφτόμαστε την αποτελεσματικότητα μιας πολιτικής κυρώσεων. Αυτό είναι άλλωστε και το ε, περιεχόμενο της έκθεσης της κυρίας Πορτέλα, την οποία βρήκα ιδιαίτερα σημαντική, και προτείνατε ο ρόλος των επικεφαλής των αποστολών ε, στις ε, χώρες μέλη είναι πολύ σημαντικός. Ε, συμφωνώ απολύτως και ίσως θα έπρεπε να το εγγράψουμε και αυτό στην έκθεση. Ζητώ συγγνώμη στον κύριο Σαλαβράκο και στον κύριο Κούκαν, διότι δεν μπορώ να απαντήσω στη γλώσσα τους. Δυστυχώς μέχρι εδώ φτάνει η γνώση μου στην περίπτωση αυτή, αλλά Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κύριο Σαλαβράκο, διότι μένει στον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών, γεγονός που κατ' εμέ είναι μία από τις ουσιώδεις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στη συγκεκριμένη συζήτηση. Ε, στον κύριο Κούκαν, για την ανησυχία του για την ανάγκη για ένα συγκεκριμένο ορισμό και την ανάγκη να απαντούμε με ευελιξία. Κύριε Κούκαν, ε, είχατε κι εσείς ε, ανάλογες θέσεις όπου χρειάστηκε να απαντήσετε με αυτόν τον τρόπο και χαίρομαι ιδιαίτερα ε, διότι μας δίνετε τη γνώση σας στο θέμα αυτό. Κύριε Ζάλα, εσείς πολύ ευγενικά κάνατε τρεις σημαντικές παρατηρήσεις στην έκθεση όχι μόνο για το γεγονό ότι δεν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ κρατών μελών, αλλά ε, ότι θα πρέπει να ε, θυμούμαστε την συναλλαγή που γίνεται μεταξύ κυρώσεων και δημοκρατικών μέτρων. Και αυτό κάπου θα πρέπει να το συμπεριλάβουμε στην έκθεση. Αναφερθήκατε επίσης ε, το, στο θέμα των παιδιών των ε, ηγετών που αποτελούν στόχο. Υπάρχει μια συγκεκριμένη υπόθεση που βρίσκεται ενώπιον του ε, Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για το γιο ενός επιχειρηματία από την Μιανμάρ που βρίσκεται υπόθεση που είναι ανοιχτή αυτή τη στιγμή και εκεί θα πρέπει να το εξετάσουμε το ζήτημα. Ίσως χρειάζεται περισσότερη συνοχή να έχουμε διάφορα μέτρα πολιτικής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε με τους επικεφαλείς ε, αυταρχικών καθεστώτων. Κύριε Κέλα, κύριε Πάσκου, ε, και οι δύο αναφερθήκατε στα προβλήματα ορισμών, όπως και κάποιοι άλλοι, και ο κύριος Κασουλίδης αναφέρθηκε στη σημασία ενός ε, κώδικα διοντολογίας ε, πριν ε, συμβεί το οτιδήποτε. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση, ο κώδικας διοντολογίας μπορεί να είναι και ιδιαίτερα σημαντικός. Δυστυχώς όμως η πείρα μου είναι ότι τηρούνται κυρίως στην παραβίασή τους και θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να ενισχύσουμε τη συζήτηση στην κοινωνία για το πώς αυτοί οι κώδικες δεοντολογίας εφαρμόζονται στην πράξη. Κύριε Πάσκου, εσείς αναφερθήκατε στην ανάγκη ευελιξίας και πάλι και στην ανάγκη να εξεύρουμε την κατάλληλη ισορροπία στην έκθεση μεταξύ ελαστικότητας και αρεχών. Και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι αρχές μπορούν να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο. Η κυρία Γέγκλε στην παρέμβασή της ρώτησε τι ρόλο μπορεί να ε, διαδραματίσει το Κοινοβούλιο στον ορισμό και την εποπτεία της πολιτικής ελπίζω ότι ένα από τα ωφέλη αυτής της έκθεσης θα είναι ακριβώς ότι θα αρχίσουμε να εξετάζουμε τι ρόλο μπορούμε να διαδραματίσουμε για τον καθορισμό και την εποπτεία της πολιτικής μας και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις εξουσίες που μας δίνονται μέσω της συνθήκης της Λισαβόνας στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ λοιπόν κύριε Πρόεδρε όλους όσους παρενέβησαν. Προσβλέπω σε ε, περαιτέρω συζητήσεις επί του θέματος και θα λάβω υπόψη μου φυσικά και σχετικές τροπολογίες που θα υποβληθούν και ε, εν ώψη της συζήτησης θα καταθέσω και εγώ τροπολογίες οι οποίες ελπίζω ότι θα βοηθήσουν να έχουμε μια έκθεση με ευρύτερη συνένεση στην Επιτροπή. Θα έλεγα πριν δώσω το λόγο στην ε, κυρία Πορτέλα ότι ο κύριος ε, Σαρουσβόλκη ε, είναι ένας καλός ανταγωνιστής για σας γιατί μας εντοπωσιάσατε, αλλάξατε τόσες γλώσσες. Παρακαλώ κυρία Πορτέλα. Η κυρία Γέγλε έθεσε ένα σημαντικό ερώτημα, δηλαδή τι ρόλο μπορεί να παίξει το Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο συχνά ζητάει να επιληθούν κυρώσεις έναντι τρίτων χωρών και αυτό το οποίο ζητείτε τώρα είναι να ασκήσει και τον ίδιο ρόλο στον, στην επιβολή αυτών των κυρώσεων. Δηλαδή γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε περιορισμό ταξιδιού αλλά όχι εμπάργο όπλων ή γιατί εμπάργο όπλων και όχι οικονομικές κυρώσεις. Και γιατί μπήκε κάποιος σε μια μαύρη λίστα ε, και γιατί όχι. Και πόσο πιστική είναι η εξήγηση του Συμβουλίου. Εδώ πέρα μπορεί να παίξει κεντρικό ρόλο το Κοινοβούλιο. Δεν ξέρω αν έχετε την εκθεσή μου πρόχειρη. Ακριβώ αυτά τα σημεία έχω αναφέρει στι συστάσεις υπαριθμών 6 και 7. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας υπενθυμίσω πως η προθεσμία για τις ε, τροπολογίες είναι στις 17 Οκτωβρίου σε 6 ώρα το απόγευμα και η συζήτηση θα είναι στις 22 Νοεμβρίου. Επόμενη συνεδρίαση 11 Οκτωβρίου. Ολόκληρη τη μέρα θα έχουμε τον πρόεδρο της ΚΝΕΣΕΤ και τον προεδρεύοντα της Ελβετικής Συνομοσπονδίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.